συνάδελφοι. Allez, Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, παρακαλώ. Και να ξεκινήσουμε από το σημείο την απόφαση που θεσπίζει το δικό πρόγραμμα υλοποίησης προγράμματος Horizon Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Ήτρε και θέλω να στήσω την προσοχή σας ότι ταυτόχρονα θα συζητήσουμε δύο γνωμοδοτήσεις. Η μία αφορά την πρόταση κανονισμού που θεσπίζει το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη και το άλλο αφορά την απόφαση που θεσπίζει το ειδικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα το σκέλος των μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Βιρκούνεν και κατόπιν θα κάνουμε μία συζήτηση και θα ζητήσουμε και την ε, γνώμη της Κομισιόν. Καταρχήν, η κυρία Βιρκούνεν. Όταν είστε έτοιμοι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε τον ορίζοντα Ευρώπη και την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την Επιτροπή Ήτρε. Χθες μόλις οι συντονιστές επιβεβαίωσαν το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση στις 15 Νοεμβρίου. Θα έχουμε λοιπόν λίγο παραπάνω από ένα μήνα για να δουλέψουμε πάνω στη γνωμοδότηση. Σε δύο δηλαδή γνωμοδοτήσεις, τις οποίες θα συνδυάσουμε βέβαια, παρά το ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές αποφάσεις. Την απόφαση για τον ορίζοντα, και τι 200 ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί γι' αυτό και τον κανονισμό για τον ορίζοντα Ευρώπη με λίγο πάνω από 100 τροπολογίες. Και το πιο σημαντικό φυσικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο προπολογισμό. Τι προϋπολογισμό θα έχει ορίζοντας Ευρώπη. Την Άνοιξη, αν θυμάστε, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός κατά 50% και πολλοί ευρωβουλευτές τροποποίησαν αυτήν την πρόταση, θέλουν παραπάνω αύξηση. Η δική μου πρόταση είναι αύξηση 50% όπως αποφάσισε το Κοινοβούλιο την Άνοιξη. Και αυτό θα είναι αφορμή για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την ομάδα, με τους κοιόδες εισηγητές, πώς δηλαδή θα καταρτιστεί ο προπολογισμό. Βέβαια πρέπει να συντονιστούμε και με την Επιτροπή Ήτρε και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, αλλά θα κάνουμε και τη δική μας πρόταση για το πώς θα χωρίσουμε τα κονδύλια αυτά σε τομείς. Βέβαια, ο τομέας των μεταφορών χρειάζεται χρηματοδότηση για πολλούς λόγους, επίσης, η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι το 35% των κονδυλίων θα διατεθεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για έρευνα και ανάπτυξη στον χώρο των μεταφορών, αποδέσμευση από χρήση άνθρακα. Νομίζω πως αυτός ο τομέας θα είναι από τους πιο σημαντικούς φαίνεται και από τις τροπολογίες άλλωστε, και αρκετά μέλη αναγνωρίζουν το γεγονός ότι ο τουρισμός δεν είναι ορατό στην πρόταση της Επιτροπής όσο θα έπρεπε. Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ευρώπη με μεγάλες προοπτικές και η έρευνα και η ανάπτυξη χρειάζεται και στον τομέα λοιπόν του τουρισμού, όχι μόνο στις μεταφορές. Επίσης, θεωρώ πως πολύ σημαντική θα είναι και η συζήτηση για το γραφειοκρατικό φόρτο Το βλέπουμε κιόλα αν προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Και θα διευκολύνει τόσο την ε, Κομισιόν όσο και τους ε, διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς αν ε, μειωνόταν η γραφειοκρατία. Νομίζω πως τη γνωμοδότηση πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Επίσης, γνωρίζουμε πως από όλα τα κράτη-μέλη κάποια υποφελούνται περισσότερο από τον ορίζοντα Ευρώπη με πολύ θετικά αποτελέσματα και άλλα τα οποία υστερούν. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη και τους φορείς τους για να συμμετέχουν περισσότερο στο μέλλον, στα προγράμματα αυτά και στον ορίζοντα Ευρώπη θα είναι πολύ σημαντικό οι δράσεις να βασίζονται στην αριστεία και να παρέχονται περισσότερες δυνατότητες σε χώρες, φορείς και συμμετέχοντες για ενισχυμένη συμμετοχή. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις τροπολογίες σας. Αναμένω τη συνάντηση των σκιωδών. Στείλαμε μόλις τις ε, τροπολογίες για μετάφραση και λάβαμε ήδη τις μεταφράσεις. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δουλειά πάνω στους συμβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερκούλα. Έχω τώρα την ευχαρίστηση να υποδεκτώ στην Επιτροπή μας όλα τα μέλη του σχεδίου Εμετράκη. Αν δεν χωράτε, μπορείτε να καθίσετε και στις θέσεις που είναι πιο μπροστά. Είστε πρόσδεκτοι. Καλώς ήλθατε. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε τις αντιπροσωπείες ε, του Μαρόκου, της ε, Τινησίας, ε, της Ιορδανίας, του Ισραήλ που εργάζονται για αυτό το project για τη συνεργασία Ευρώπης και Βορειός Αφρικής. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή των Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορούμε να τους χειροκροτήσουμε για να τους αποδεχτούμε όπως πρέπει. Λοιπόν, είμαστε σε εξέλιξη στις εργασίες μας. Συζητούμε την έκθεση της κυρίας Βερκούνεν για ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο λέγεται Horizon Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα θέσει σε εφαρμογή ένα πολύ σημαντικό πεδίο δράσεων, γιατί καλύπτει το κλίμα, την ενέργεια, την κινητικότητα, τις μεταφορές και τι θα κάνουμε στο μέλλον έτσι ώστε οι διασυνδέσεις ε, να μπορούν ε, να λάβουν χώρα και να χρηματοδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν βάσει πιλωτικών σχεδίων. Λοιπόν, είστε ευπρόσδεκτοι, εμείς συνεχίζουμε τη συζήτηση μας και θα δώσω το λόγο στην κυρία Πλούση εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εμείς ε, στηρίζουμε τη γραμμή που επέλεξε η συγγήτρια. Έχω την ευρεία στήριξη της ομάδας μου σε αρκετά σημεία. Ορισμένα από αυτά έχουν ως εξή. Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε προς την απλούστευση του ορίζοντα Ευρώπη και να δώσουμε έμφαση στην αριστεία. Αυτό θα γίνει κυρίως μέσω απλούστευσης της, γραφή, της διοικητικής διαδικασίας, η οποία θα βοηθήσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην ισότητα των φίλων και στην ε, ίση εκπροσώπηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσφέρονται αντίστοιχα προγράμματα. Προτείνουμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ιδιαίτερα για τον τομέα των μεταφορών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα... τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν, χρειάζεται να θεσπιστούν κριτήρια προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ε, μετά, πρέπει να προστατεύονται τα εμπορικά μυστικά από περιπτώσεις ε, κατάχρησης πέρα από τα προσωπικά δεδομένα. Δυστυχώς ε, δεν έχουν όλες οι χώρες εταίροι μας ικανοποιητικά πρότυπα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας των εμπορικών μυστικών. Πρέπει επίσης ε, να διευκρινιστεί με περισσότερη σαφήνεια η συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Είμαι σίγουρη πως με την εισηγήτρια θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και θα οδηγηθούμε σε εξίσου καλές συμβαστικέ προτάσεις. Ελπίζω η Επιτροπή Μεταφορών να παρουσιαστεί αποφασισμένη και να καταρτήσει μια υποδειγματική γνωμοδότηση στην, ε, για την Επιτροπή Ήτρε. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριε Κύριε Μάισνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων, ήθελα να πω ότι έχουμε περίπου την ίδια γραμμή ε, σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση. Σίγουρα και εμείς θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία, το διοικητικό άχθο, θέλουμε αριστεία στις επιστήμες και έμφαση σε αυτό έμφαση στην ε, ηγεσία στη βιομηχανία και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για ε, να ωφεληθεί η καινοτομία και η έρευνα. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Και η άλλη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η θάλασσα, οπότε Αυτή την ε, αγάπη μου την έχω μεταφέρει και στο ε, Cluster Food and Resources. Συμπεριλαμβάνεται και η θάλασσα και η ναυτιλία και η αλληλεία. Διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε αναφορά στην αλληλεία και την ε, πολιτική για τη θάλασσα. Προσπάθησα λοιπόν όπου μπορούσα να εισαγάγω και αναφορές σε αυτά. Επίση, ζήτησα αύξηση για αυτή την ομάδα από 10 δισεκατομμύρια σε 16. Τρόφιμα λοιπόν, φυσική πόρη, θάλασσες και ωκεανή. Σε αυτήν την ομάδα έχω υποβάλει πρόταση για να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Αυτά ε, εν ολίγης από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε ο κύριος Νταλούντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χτες ε, η εξέδωσε μία έκθεση ε, που την υπέγραψαν κορυφαίοι επιστήμονες σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Ο δημοσιογράφος του BBC συνόψισε την έκθεση με ένα μήνυμα τριών λέξεων από τους επιστήμονες τους πολιτικούς. Δράστε τώρα, ηλίθιοι. Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και να επηρεάσουμε το έργο μας με τον οριζόντα Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό στην καινοτομία και στην έρευνα, να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις αλλαγέ που είναι αναπόφευκτες. Στο προηγούμενο πρόγραμμα Horizon 2020 είχαμε δεσμεύσει πόρου για ε, project σχετικά με την κλιματική αλλαγή, όμως ε, στην ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου χάσαμε το στόχο όπως φάνηκε για 5%. Επίσης, ε, τώρα όλα τα προγράμματα συνσέφεραν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Καταρχήν, να αυξήσουμε ουσιαστικά τη δέσμευση πόρων ε, για τα κλιματικά project στο 50%. Δεύτερον, ισχυρότερη νομοθεσία για να πετύχουμε τους στόχους. Και τρίτον, να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κλιματικά προγράμματα συνεισφέρουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή να μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε σε αυτή. Αυτό πρέπει να το κάνουμε για να κάνουμε τον ορίζον, το ορίζον Ευρώπη να ε, απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό του και να μπορούμε να σεβαστούμε και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Ευχαριστούμε κύριε Ντελούντε. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή την Επιτροπή δεν υπάρχουν ηλίθιοι. σε σχέση με τον δημοσιογράφο το BBC που είπε ότι πρέπει να δράσετε τώρα η Στην ε, επιτροπή αυτή έχουμε μόνο υπεύθυνου ανθρώπους ε, και έχουμε κατανοήσει ότι καθόμαστε πάνω σε ένα ηφαίστειο και ότι για την κλιματική αλλαγή θα δράσουμε έτσι ώστε να αποτελέσει η προτεραιότητά μα και να είναι εγκάρσια σε όλα τα προγράμματα. Κυρία Κιλούνα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ και την κυρία Βερκούνεν. Οι ιδέες σας και οι ρεαλιστικές σας ε, προτάσεις μου αρέσουν πάρα πολύ ως Φιλανδοί βουλευτή. Νομίζω ότι η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών είναι το ζήτημα κλειδί, ιδίω όταν μιλάμε για τη μεταβολή του κλίματος ε, και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τη Συμφωνία των Περισσίων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης. Αυτό που με ανησυχεί κάπως είναι ότι συνήθως με αυτά τα προγράμματα οι μικρές και μισές επιχειρήσεις δεν έχουν πολύ καλή πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα. Και η ιδέα να έχουμε χαμηλό γραφειοκρατικό άχθος θα τους βοηθούσε βεβαίως. Αν μπορούσαν να λάβουν λοιπόν περισσότερη υποστήριξη και βοήθεια για να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν τις ιδέες τους με τις άλλες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν κάτι καλό. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα να συνδέσουμε διάφορους τρόπους μεταφοράς και διάφορα ιδιαιτεριών και να έχουμε την πολυτροπικότητα την οποία έχουμε αναφέρει πολλά και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα δεν λειτουργεί, ελπίζω κάποτε. Και να κάνουμε κάτι παραπάνω για να την προωθήσουμε. Επίση, όταν ε, μιλώ για εταιρικέ σχέσεις, για τη δυνατότητα διασύνδεσης διαφορών πραγμάτων, Εδώ σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο με την κυρία Μάισνερ. Να συνδέσουμε λοιπόν τα τρόφιμα, το νερό, τις μεταφορές, όλους τους κλάδους να τους συνδέσουμε και μετά να έχουμε αλλαγές στην οικονομία μας και στα συστήματά μας. Έτσι ώστε να εντάξουμε σε αυτό και την προοπτική του κλίματος. Αυτά είναι τα σύντομα σχολιά μου και ανυπομονώ να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κιλόνεν. Θα στραφώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιο είναι το σχέδιο δράση και το φύλλο για αυτό το πρόγραμμα ορίζοντα 2020. Η κυρία Ρομπέρτα Ζόμπι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που δίνεται στην Κομισιόν την ευκαιρία να σχολιάσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με την Επιτροπή σας. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα που θέσατε που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για μας. Και πιστεύω ότι δικαιοδοτήσετε ορθά στην πρόταση της Κομισιόν. Αναφέρομαι στους στόχους της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, το κλάστερ ε, του κλίματος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Έχουμε εδώ μια συστημική προσέγγιση για να πετύχουμε αυτό το στόχο και τις γραμμές δράσης που προτείνονται. Όλα αυτά στοχεύουν σε μείωση των εκπομπών και της ρήπανσης γενικότερα. Ο στόχος του 50% που αναφέρθηκε είναι ένας στόχος που έχει ήδη επιτευχθεί από το πρόγραμμα μεταφορών και το πρόγραμμα ενέργειας στον ορίζοντα 2020. πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν καλά προγράμματα που δεν σχετίζονται τόσο πολύ με το κλίμα, όπως ε, το ΕΛΤΣ, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία, λαμβάνοντα υπόψη ότι και το πρόγραμμα Horizon 2020 καλύπτει κλάδους που δεν είναι τόσο σχετικοί, δεν έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο προς το κλίμα. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζεται ορθά και σημειώνουμε την πρόταση να κάνουμε ένα συνδεσμό μεταξύ της κινητικότητας ε, στη μεταφορές και στον τουρισμό, πιο ξεκάθαρο, σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Η πρόθεση της Κομισιόν είναι να προωθήσει αυτά τα οποία είχαμε ήδη ξεκινήσει στον ορίζοντα 2020 και να απλουστεύσουμε περισσότερο την συμμετοχή και την πρόσβαση. Αναφέρθηκε και το θέμα της διεύρυνσης, νομίζω και αυτό είναι σημαντικό Προσπαθούμε να βρούμε την ορθή ισορροπία στην πρότασή μας μεταξύ της ανάγκης να διασφαλίσουμε την αριστεία, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε ορθά το κενό συμμετοχής των κρατών μελών. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα συνεχίσουμε τις ε, εργασίες με τους Σκιώδης και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή πιθανότητα να υπάρξει μια καλή γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουμε να επικεντρωθούμε στους ίδιου στόχους. Η έκθεση θα είναι πολύ καλή, λοιπόν, που θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο το Νοέμβριο. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και σας ευχαριστώ όλους ε, για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστούμε κύριε Βερκούν. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι την 3η 11 Σεπτεμβρίου λέει η Πρόεδρος. Στι 3 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με την πρόταση κανονισμού σε σχέση με τις απαιτήσει έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων σε ό,τι αφορά την γενική της ασφάλεια και την προστασία επιβατών των οχημάτων και το βάλλον των χρηστών του, της οδού. Είναι μια έκθεση προ την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ο κύριο Βαν Μίντελμπρουκ είναι ο συγητή. Καλημέρα σα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η βελτίωση της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές είναι μία από τις βασικές προκλήσεις όχι μόνο της Επιτροπής αλλά και του υποφαινόμενου. Γι' αυτό υποβάλλουμε μία γνωμοδότηση στην ΙΜΚΟ για την ασφάλεια στις ε, οδικές μεταφορές. Ο κύριος Κόχ είχε μία προγενέστερη έκθεση για την ασφάλεια των ε, οχημάτων. Μας ενδιαφέρει ο τύπος ε, ε, ασφάλειας γιατί μας απασχολούν τα θανατηφόρα και γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχέα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μεγάλη επίπτωση και αντίκτυπος για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές και για να αποτραπούν τα ανθρώπινα λάθη. Το θέμα της ταχύτητας, η αναγνώριση, το σύστημα ώστε να κρατάμε τη λωρίδα μας, καθώς και τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται. Επίσης, αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει και την αυτοκινητοβιομηχανία και για την αυτόνομη οδήγηση θα ήθελα να υπογραμμίσω διάφορα σημεία τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν. Η ασφάλεια θα πρέπει να εγγυάται σε ολόκληρη την Ευρώπη για όλα τα οχήματα, χωρίς να έχει σημασία ο τύπος οχήματος ή το πόσο πολυτελές όχημα είναι. Θα πρέπει να αφορά όλα τα οχήματα. Επίσης, η επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να εντάσσεται στον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν περισσότερες ε, εγγυήσεις, ιδιαίτερα ως προς την καταγραφή συμβάντων και μέσα στα πλαίσια της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης στα στοιχεία. Τα στοιχεία ασφάλειας επίσης που θα πρέπει να δοκιμαστούν πριν από την εφαρμογή. Για παράδειγμα, το θέμα της ε, βοήθειας ε, κατά την προσπέραση θα πρέπει να ε, αφορά το γεγονός ότι ο οδηγός θα πρέπει να έχει μία βοήθεια. Επίσης, η σηματοδότηση, η οδική σηματοδότηση είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη σχέση κόστους ωφελίας, δηλαδή θα πρέπει τα οχήματα να είναι προσβάσιμα για τον τελικό ε, χρήστη. Τα στοιχεία ασφάλειας θα πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη και γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι χρήστες να προωθήσουν την ασφάλεια αυτή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσμένω να συνεργαστούμε με τους άλλους σκιώδεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Εύα Μίλτενμπεργκ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόρ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Φων Μίλτενμπουργκ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ καλή γνωμοδότηση, η οποία αποτελεί μια εξίσου καλή βάση για την επόμενη φάση. Βέβαια, δεν ήσασταν φιλόδοξο, δεν έπρεπε όμω και να είστε. Και νομίζω πω αυτό έχει να κάνει με το ότι είστε ικανοποιημένο από την πρόταση τη Κομισιόν. Συμμερίζομαι την ε, ικανοποίησή σα, γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι σχεδόν όλες οι προτάσεις ε, που είχα κάνει στη δική μου έκθεση για την ασφάλεια ε, και την προστασία της ανθρώπινης ζωής έχουν ληφθεί υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στην άποψη, στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω πως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και πρέπει να φροντίσουμε να συνεχίσουμε ενωμένοι έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην δημιουργία νέων συστημάτων βοήθεια στα οχήματα έτσι ώστε να βελτιώσουν την ε, ασφάλεια της οδήγησης χωρίς ε, ταυτόχρονα να αυξήσουν κατά πολύ το κόστος. Έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τους ε, κινδύνους και τους προβληματικούς τομείς. Και έχουμε αναγνωρίσει το ότι δεν πρέπει τα συστήματα βοήθεια στην οδήγηση να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους. Τα συστήματα αυτά τα οποία αναφέρατε θα πρέπει φυσικά να έχουν ως κύριο προτεραιότητα την ασφάλεια των οδηγών και να συνοδεύονται από ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι ε, να έχουν ως γνώμονα το κόστος. Γι' αυτό θεωρώ ότι επιδέχεται βελτιώσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να καταλήξει σε μια πραγματικά υποδειγματική, εξαιρετική πρόταση. Πέρυσι είχαμε 35.000 βαριά τραυματίες σε, σε τροχαία ατυχήματα και περίπου 15.000 νεκρούς. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια και επίσης να ε, μην παραμελούμε τον συνοδηγό. Θα υποβάλω τροπολογίες έτσι ώστε να κατεργαστούμε ακόμα περισσότερο αυτό το ήδη κατεργασμένο διαμάντι που μας ε, παρουσίασε η Επιτροπή, οι οποίες θα αφορούν τα συστήματα ελέγχου και συστήματα υποβοηθούμενη οδήγηση τα οποία θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε. Θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσει σχετικά με αυτό και θα πρέπει να ε, θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα. Μετά, ποια συστήματα θα μπορεί να ελέγχει ο οδηγός. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις εδώ υπάρχουν ορισμένα συστήματα τα οποία βοηθούν να, να παρακάμψει κάποιος την κίνηση στο δρόμο και κάποια άλλα ε, τα οποία αφορούν την ίδια την οδική ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ε, βάση στις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Σε σχέση με τα ερωτήματα που εθίγησαν από τον εισηγητή για αυτά τα συστήματα συνδρομής, θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό ατυχημάτων και τον αριθμό των τραυματιών και να αντιμετωπίσουμε το ανθρώπινο λάθος. Σε σχέση με τον κανονισμό της Επιτροπής εμπεριέχει στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων για να μειωθούν τα ανθρώπινα λάθη που μπορούν να ε, οδηγήσουν σε ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι και θανατηφόρα. Θα πρέπει λοιπόν ο οδηγός να δεχτεί αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας και να έχει και όλες τις πληροφορίες για την ενδεχόμενη ε, συνδρομή κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει αυτό το στοιχείο να ληφθεί υπόψη, γιατί όταν υπάρχουν συστήματα, ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Γιατί καμιά φορά όταν οι υποδομές αυτές δεν συντηρούνται, τότε ε, ανακύπτουν ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και στοιχεία συνδρομής προς τον οδηγό και χαίρομαι για τη συνεργασία μεταξύ όλων των συναδέλφων ε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία καλή και φιλόδοξη γνωμοδότηση με βάση και την περσινή γνωμοδότηση που είχαμε για να βελτιώσουμε αυτή την ε, πολύ καλή σχέση που είχαμε και με τον προγενέστερο κανονισμό. Η κυρία Κιλόνεν έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε Ματής για, αυτή το, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και φυσικά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση έχει γίνει πολύ σοβαρή εργασία και θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα με την ασφάλεια. Παράλληλα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κινητικότητα των εκπομπών, δηλαδή να υπάρχει ε, συνάρτηση ασφάλειας και εκπομπών και αυτό μας απασχολεί είναι και η αυτόνομη οδήγηση που φαίνεται ότι προσεγγίζει όλους τους τρόπους μεταφορών, αλλά ιδιαίτερα τις οδικές μεταφορές και τις θαλάσσιες. Τα συστήματα όταν είναι εύχριστα και όταν δεν φοβάται ο άνθρωπος, έχει δηλαδή όλες τις πληροφορίες και τις χρησιμοποιεί σωστά, τότε ε, φτάνουμε σε καλό αποτέλεσμα. Όμως έχουμε τα ε, συστήματα TBS, όπου όταν δεν έχει το αυτοκίνητο διαδίκτυο μπορεί να στείλει τις πληροφορίες. Άρα έχουμε τα παλαιά συστήματα και τις, ε, τον παλιό εξοπλισμό. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι εύχριστες αυτές οι πληροφορίες. Ας συνεχίσουμε με την πολύ καλή εργασία. Πιστεύω ότι θα δώσουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση στην ΙΜΚΟ, η οποία θα την εντάξει στις δικές της εργασίες. Θα ήθελα τώρα να λάβω και εγώ το λόγο γιατί όλοι θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Γιατί τα αριθμητικά στοιχεία μας πληγώνουν 25.000, 25.000, 26.000 πλέον, 26.000 θανάτους στη, στα οδικά δίκτυα κάθε χρόνο ένας θάνατος αντιστοιχεί σε επτά τραυματίες, τραυματίες που μένουν ε, ανάπηροι στην ουσία. Πολύ ψηλό το ποσοστό λοιπόν. Άρα θα πρέπει να αντιδράσουμε και να προβάλλουμε περισσότερα μέτρα γιατί θα πρέπει να φτάσουμε στον ευκταίο στόχο, μηδενικό ποσοστό θανάτων. Έχουμε την πρώτη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Κορ σε αυτό το θέμα, αλλά όταν ε, μιλάμε για οδική ασφάλεια θα πρέπει να έχουμε μία ολιστική θεώρηση. Εξαρτάται από το όχημα, από τις υποδομές, από τον οδηγό, αλλά και από όλα τα μέτρα ασφάλειας, ενεργητικής και παθητικής σε όλα τα επίπεδα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τακτικούς ελέγχους στα οδικά δίκτυα, διότι η βασική αιτία θανάτου ξέρουμε η μια σοβαρή αιτία είναι η ταχύτητα, η υπερβολική ταχύτητα κυρίως. Και υπάρχουν χώρες που λαμβάνουν μέτρα. Η Γαλλία έχει επανεισαγάγει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα σε ορισμένες διαδρομές. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Κόρ στην έκθεσή του, θα πρέπει να ε, ορίσουμε ποσοστιες ε, αναλογίες ελέγχου οχημάτων κατηγορίας M1 και N1 και μιλώ για αυστηρούς ελέγχους όταν δούμε τον υποχρεωτικό χρόνο εργασίας και το χρόνο ανάπαυσης για τα βαρέα οχήματα, κάτι που ξεχνάμε στις εκθέσεις, θα είναι άλλοι οι συσχετισμοί και θα πρέπει να έχουμε ε, διάβλους, ε, διόδους πρόσβασης για τα οχήματα, λωρίδες έκτακτης ανάγκης δηλαδή, καθώς και μέτρα ασφάλειας για την ε, ηλεκτρική κινητικότητα. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο σκέλος του έργου μας. Θεωρώ ότι σήμερα υπάρχει η τεχνολογία, το είπατε και εσείς, ε, κυρία Κιλόνεν, και εσείς, κύριε Βαν Μίτελμπεργκ. Το αναφέρατε. Μιλάμε για την ψηφιακή επανάσταση η οποία θα πρέπει να μας οδηγήσει σε πρόβλεψη. Ο κύριος Βιν Βαντεκάμπ Κάμπ, θα ασχοληθεί με την έκθεση για τα αυτόνομα οχήματα και θα πρέπει να διευθετήσουμε και αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ασφάλεια αν δεν μιλάμε και για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αν δεν έχουμε ένα σχέδιο για τα open data. Και εάν δεν μιλήσουμε για ευθύνη και για κυρώσεις, ποιος είναι υπεύθυνος στη χρήση των οδικών δικτύων και ως προς την ψηφιακή επανάσταση θα πρέπει να επεκτείνουμε και το σύστημα e-call που διαθέτουν ορισμένα οχήματα ήδη σήμερα Θα ήθελα όμως να υπάρχει και στα βαρέα οχήματα, τα λεωφορεία, ε, τα τουριστικά λεωφορεία και τα βαρέα οχήματα. Και αυτό αφορά και θέματα που σχετίζονται με την χρήση της ζώνης ασφαλείας καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούν εγκλωβισμό. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και σύστημα ανείχνευσης κινδύνου να αποκοιμηθεί κανείς στο τιμόνι. Έχετε δίκιο κύριε Βαν Μίτελμπουργκ. Θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη οδική σήμανση και ιδιαίτερα σήμανση στην άσφαλτο. Και θα πρέπει να βρούμε και ευφύη συστήματα για να μπορέσουμε να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα, η σήμανση stop και πολλές φορές η σήμανση γενικά οδηγεί σε λάθη, είναι λυπής. Άρα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους στην οδική ασφάλεια και αυτό το μαθαίνει κανείς από μικρός. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τους κινδύνους ε, των οδικών δικτύων για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίσουν. Τώρα, θα ήθελα η Ντέζε η Γενική Διευθυντή Γκρό και ο κύριος Οσίν να μας μιλήσει για το τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Thank you very much. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις σας. Η Κομισιόν θέλει να τονίσει ότι ακολουθώντας και πολλές από τις συστάσεις της έκθεσης ΚΟΧ αυτή ήταν ένα από τα κύρια στοιχεία που άφησε την Κομισιόν στο να εκπονήσει αυτή τη φιλόδοξη πρόταση. Όντω βασίζεται κυρίως στην τεχνολογία και στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τον παράγοντα του ανθρωπίνου λάθους, αλλά όχι και μόνο. Αλλά εισαγάγει και κάποια μέτρα κοινή λογική, όπως θα το αποκαλούσα. Και θα ήθελα να αναφέρω την πρόταση να έχουμε ε, ουσιαστικά άμεση, ε, απέτηση άμεσης ε, όρεσης για τα φορτηγά. Ε, έχουμε για τα φορτηγά απέτηση μόνο να υπάρχουν καθρέφτες, έμεσης όρεσης δηλαδή. Έτσι λοιπόν, Θέλουμε τώρα με τα μέτρα αυτά να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως τους ποδηλάτες και τους πεζούς και με το νέο σχεδιασμό της καμπίνας των φορτηγών θα μπορέσουμε ο οδηγός μάλλον, θα μπορέσει να έχει πολύ πιο άμεση όρεση, δηλαδή είτε ε, επαφή, ε, κατευθείαν ε, επαφή όρεσης με τους πεζούς και τους ποδηλάτες και αυτό φυσικά μπορεί να σώσει πολλές ζωές. Τέθηκαν πάρα πολλά σημεία. Αλλά να πω ότι συμφωνούμε μας υπόθηκαν. Βεβαίω, σε σχέση με την καταγραφή των δεδομένων. Ακούσαμε τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, για το πόρτο των δεδομένων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τη χρήση αυτού του καταγραφέα δεδομένων μόνο στην ανάλυση δεδομένων. Και φυσικά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων θα ισχύει εδώ. Επίσης θα υποστηρίξουμε κάθε πρόταση να τελειοποιήσουμε περαιτέρω τη διατύπωση προκειμένου να δώσουμε ασφάλεια ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Φυσικά θα πρέπει να βρούμε και μια κατάλληλη ισορροπία. Ίσως ε, να μην βάλουμε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες στον κανονισμό, γιατί οι λεπτομέρειες ε, θα ρυθμιστούν στη δευτερογενή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμη περισσότερο η αρχή σε ό,τι φορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως ε, παραδείγματο χάρη το Intelligence Speed Assistance, αυτή η βοήθεια. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι μπορεί να μην είναι απολύτως αξιόπιστο και η αξιοπιστία αυτού του συστήματος εξαρτάται πάρα πολύ από την σήμανση την οδική και από τους ψηφιακούς χάρτες που μπορεί να μην είναι πάντοτε επικαιροποιημένη. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που η Κομισιόν δεν προτείνει ε, το σύστημα αυτό ε, να παρακαμφθεί. Δηλαδή, θα μπορεί ο οδηγός να παρακάμπτει το σύστημα αυτό αν θεωρεί ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει δεν είναι σωστές ή θα αποφασίσει, συνειδητά όμως, για οποιοδήποτε λόγο, να οδηγήσει πάνω από το όριο ταχύτητας. Το κάναμε αυτό γιατί δεν έχουμε τη διασφάλιση ότι το σύστημα θα είναι 100% αξιόπιστο. Και επίσης για να δείξουμε στον οδηγό ότι πρέπει να κερδίσει την ε, αποδοχή του συστήματος. Δηλαδή, αν έχεις ένα σύστημα που πάντα κάνει μπιπ, δεν μπορείς να προσπερνάς, ε, τότε ε, έχουμε ένα θέμα με την αποδοχή του συστήματος. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία και εδώ, αλλά πολύ στενά συνεργαζόμαστε στην Κομισιόν με τους συναδέλφους από τα αρμόδια τμήματα για τις μεταφορές, με τη γάμα δελτα έτσι ώστε και η πρότασή τους για τις οδικές ε, υποδομές να λαμβάνει υπόψη το θέμα της οδικής σήμανσης. Πρέπει να έχουμε μια γενική προσέγγιση. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό εδώ με το μέτρο ασφαλείας για την έγκριση τύπου και μέσω των υποδομών. Αυτά. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο εισηγητής για καταληκτικά σχόλια. Ναι, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι εύκολα θα φτάσουμε σε συμβιβασμό γιατί υπάρχει μεγάλη λογική σε αυτό που υπόθηκα. Θέλω να αναφερθώ στο τελευταίο θέμα. Και εγώ σύμφωνα με την Κομισιόν ότι πάντοτε θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο την αποδοχή των συστημάτων ε, στο ευρύτερο κοινό, αλλά και τις ε, προϋποθέσεις, τις συνθήκες που μπορεί πριν το χάρη να επιβάλλουν ε, ότι μπορεί να παρακάψουμε ένα σύστημα και πριν το χάρη του Intelligence Speed Assistance είναι ένα παράδειγμα, αν σκεφτούμε παραδείγματο χάρη τι συνέβη φέτο με τι δασικέ πυρκαγιέ, αν χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορα να εγκαταλείψει μια επικράτεια, φυσικά ε, η ασφάλεια σχετίζεται με την ευμερία τη οικογένειά σου. Βέβαια, πάντοτε αυτό υπερβαίνει την απέτηση του ρίου ταχύτητα, του σεβασμού του ρίου ταχύτητα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και κάποια λογική όταν επιβάλλουμε κάποια τέτοια συστήματα και φυσικά θα πρέπει να μπορούμε να τα παρακάμπτουμε. Εγώ νομίζω ότι όλα όσα είπαν οι σχεδεσίτες μπορούν ε, να ενταχθούν σε συμβιβασμό. Νομίζω ότι θα παραδώσουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση στην ΙΝΚΟ και εγώ είμαι και ένα πληρωματικό μέλος στην ΙΝΚΟ και θα διασφαλίσουμε ότι η γνωμοδότηση τραν θα ακουστεί. Θα εισακουστεί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σας. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι στις 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και συνεχίζουμε. Με το επόμενο σημείο, πρόταση οδηγία σε σχέση με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και καταργώντας την οδηγία του 2009-22. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ο κύριος Μέγερ, παρακαλώ, έχει το λόγο, συζητητής. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόταση ε, είναι πολύ θετική, την καλωσορίζουμε, η οποία είναι μια πρόταση που θα παρέχει προστασία στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία για τις συλλογικέ προσφυγές είναι μια έκθεση που έχει αναλάβει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Μας ζητήθηκε να καταρτήσουμε γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή και για τους ε, μηχανισμούς που την στην οδηγία. Είναι πολύ σημαντική οδηγία για τους καταναλωτές και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και λόγω της ε, επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας ε, στον χώρο της προστασίας των καταναλωτών. Έχω προτείνει ορισμένες διαγραφές, για παράδειγμα για το αν θα πρέπει να, είναι να γίνει παραδεκτή μια τέτοια συλλογική αγωγή. Θεωρώ πως αυτό θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια έγκαιρη επικαιροποίηση της ε, οδηγίας. Επίσης, να σας υπενθυμίσω την οδηγία για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, η οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας ορισμένων διαδικασιών και να οδηγηθούμε έτσι σε ε, Μετά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για ε, να οδηγούνται επιχειρήσεις σε αυθαίρετες ε, ενέργειες οι οποίες έχουν όφελος μόνο το κέρδος. Μετά, έχουμε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ πως χρειάζονται τροποποίηση και θα καταθέσω για αυτά τις ε, ανάλογες τροπολογίες. Λοιπόν, αρχίζουμε από τους ορισμούς ε, για τους ε, αρμόδιους φορείς. Χρειάζεται ακριβέστερος ορισμός, όπως επίσης και για ε, το ποιος είναι αρμόδιος για την διεκπαιρέωση των συλλογικών αυτών αγωγών. Έπειτα, στις περιπτώσεις συλλογικών αγωγών ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις. Δηλαδή, η δυνατότητα συλλογικής προσφυγής θα πρέπει να γίνεται με την συγκατάθεση του καταναλωτή και όχι ε, χωρίς αυτή. Μετά, θα πρέπει να ισχύει η αρχή της ε, ίσης αντιμετώπισης και τέλος οι αμοιβέ των ε, συνηγόρων. Νομίζω πως ε, οι αμοιβέ αυτές θα πρέπει να καθορίζονται από τις ε, αρμόδιες αρχές του κάθε κράτους μέλους. Επίσης, οι αποζημιώσεις δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος ε, της ε, ζημιάς, έτσι ώστε να μην περάσουμε στις πρακτικές που ισχύουν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα λάβετε τις τροπολογίες σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλίν, Αλή Λατίφοφ. Είσαστε πρόεδρος, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή. Merci de votre présence. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θα παρακολουθήσετε τις εργασίες μας. Επειδή έχουμε καθυστέρηση εργασία, ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο για δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση, για ε, την, ε, τις ιδέες του και, εμεί, και εμείς ε, σήμερα ψηφίσαμε έναν κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών στην Επιτροπή Μεταφορών. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός. Υπάρχουν και άλλοι παρόμοιοι κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών στον αεροπορικό τομέα και στις θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα παραρτήματα, σε ποιες οδηγίες θα πρέπει να, σε, σε ποιες οδηγίες πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός, γιατί πολλές φορές Αντί να βοηθάμε τους καταναλωτές, τους μπερδεύουμε. Δηλαδή, οι καταναλωτές μπορούν να προβάλλουν τα δικαιώματά τους έναντι των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά δεν ξέρω αν πάντα χρειάζονται συλλογικές αγωγές. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο κατάλογος των παραρτημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε ε, Μαρινέσκου, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Βέβαια, έχουμε ορισμένες ε, σημαντικές αμφιβολίες για την έκθεση. Θεωρούμε πως ε, υπάρχει περιθώριο για να γίνουν καταχρήσεις, μπορεί να οδηγηθούμε σε χάος στα νομικά συστήματα υπάρχει ο κανονισμός 261 που καλύπτει τις μεταφορές. Σήμερα ψηφίσαμε για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών και δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτό το μέα στο πεδίο εφαρμογή. Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας είναι οι ενδεχόμενες συλλογικέ αγωγές χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ενημερωθεί για το ότι συμμετέχουν σε μια τέτοια συλλογική αγωγή. Για παράδειγμα, αν κερδίσουν, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να μάθει, διότι τα ποσά θα είναι μικρά και θα παραμείνουν εντός αυτής της αρμόδιας ε, οντότητας, όποια και είναι αυτή. Εάν χάσουν βέβαια, ο καταναλωτής δεν θα έχει ιδέα για το ότι συμμετείχε σε αυτήν την ε, αγωγή και υπάρχει και το θέμα του opt-out. Μετά, ποια είναι η αρμόδια οντότητα. Είναι μη, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Μία μη κερδοσκοπική οργάνωση πρέπει να έχει μηδενικό ισολογισμό στο τέλος του οικονομικού έτους και το πρόβλημα εδώ είναι πως τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς για το τι αποτελεί μη κερδοσκοπική Οργανισμό. Θα με ενδιέφερε να δω την άποψη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Και τώρα, αυτές οι αρμόδιες οντότητες, αυτά qualified entities, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν δημόσια χρηματοδότηση. Δηλαδή, τι, ο φορολογούμενος θα πληρώνει για κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες έντονες ανησυχίε και θα με ενδιαφέρει απόψη τη Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, αλλά δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών. Κυρία Μάισνερ. Κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω στα γερμανικά γιατί θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μάιερ για την αναφορά του στα δικαιώματα των επιβατών ε, αεροπορικών μεταφορών και ευχαριστώ πολύ την κυρία Φώστερ που το ανέφερε. Και τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί μιλώ εκ μέρου του κυρίου Βαλμίλτενμπουργκ, ο οποίο έπρεπε να φύγει γιατί είχε άλλε υποχρεώσει. Ο κύριο Μίλτενμπουργκ, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα εξυγχρονίσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ω ε, σκιώδη ηγητής στην Επιτροπή ΙΜΚΟ έχω συζητήσει το θέμα και εκεί κατέστη σαφέ ότι χρειάζεται κριτική εξελόγηση της πρότασης της επιτροπή. Να τονίσω πρώτα ότι η οδηγία αυτή σκοπεύει σε ε, ελάχιστη εναρμόνιση. Έπειτα, συμφωνώ με τον εισηγητή για αυτές τις qualified entities οι οποίες ε, εγκεκριμένες οντότητες ε, χρειάζονται περισσότερες ε, διευκρινήσεις. Στο άρθρο 4, τρίτον, η απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 6 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά εξαίρεση σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό να μην γίνει ο κανόνας. Τέλος, η Δύσκολε υποθέσει που περιλαμβάνουν καταναλωτέ σε πολλά κράτη-μέλη απαιτούν καλό συντονισμό. Και το άρθρο 16 αναφέρει μεν ε, κάποια στοιχεία για τη διασυνοριακή συνεργασία. Χρειάζεται όμω καλύτερη και βελτιωμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν ε, αυτές οι περιπτώσεις. Σα ευχαριστώ πολύ και ε, εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία. Ο Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και Ευχαριστώ τον κύριο Μάιερ για την εργασία του σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Νομίζω ότι το Dieselgate και τα σκάνδαλα ακύρωσης των πτήσεων της Ryanair έδειξαν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών έτσι ώστε να ζητήσουν αποζημιώσεις από αυτές τις συλλογικές οντότητες ως προς τις διασυνοριακές ε, μεταφορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αυστηρότητα των μέτρων για λόγους διαφάνειας και δημοκρατίας θα ήθελα και τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες για τις συλλογικές αυτές αγωγές και την εξέλιξή τους και αυτό αφορά και την αποζημίωση και την επανόρθωση από, τους, από τις συγκεκριμένες οντότητες. Επίσης, η πράσινη θα ήθελα να συμπεριληφθεί και να συμπεριληφθούν και οι πλατφόρμες online καθώς και τα θύματα περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Θα ήθελα λοιπόν Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε μία καρποφόρα συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ, η κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Κιθ Τέιλορ ήδη είπε αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Είμαι υπέρ μιας ισχυρότερης προστασίας για τους καταναλωτές, έστω και αν αυτό συνεπάγεται αντιπροσωπευτικές συλλογικές αγωγές. Είδαμε και με το Dieselgate ότι η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική στην Ευρώπη από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε και οι καταναλωτές στις Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ε, καλύτερη προστασία από τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε δουλειά πάνω στο σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο εισηγητή Μάιερ. Ευχαριστώ κυρία Κιλόνεν και αμέσως να δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Πιμ Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα τι είπε η κυρία Φώστερ και έκαναν μεγαλύτερη επίχυση σε μένα από ό,τι τα λόγια του κυρίου Μαρινέσκου. Στο Εθνικό Κοινοβούλιο στις κάτω χώρες εμείς είχαμε μεγάλα προβλήματα με τέτοιες αγωγές και έχω δύο ερωτήσεις ε, για τον εισηγητή. Θα πρέπει να έχεις υποστεί ζημία, πραγματική ζημία, γιατί πολύ ωραία είναι να λέμε ότι όλοι, παραδείγματος χάρη, θα λάβουν αποζημίωση όταν ε, μόνο το 10% ε, των οχημάτων της Volkswagen ε, όμως εμφάνισε προβλήματα, αλλά θα λάβουν όλοι αποζημίωση, παραδείγματος χάρη. Πολύ εξυγχρονισμένη είναι αυτή η νομοθεσία, όμως στην Ολλανδία είχαμε ε, παραδείγματο χάρη ένα πρόβλημα όπου ε, μόνο το ίμιση των καταναλών υπέστη ζημία, αλλά όλοι έλαβαν την αποζημίωση. Επομένω, τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην Κομισιόν και θα δώσω το λόγο στην κυρία Πετρέσκου. Très, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση. Νομίζω ότι πράγματι και εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την προστασία των καταναλωτών συνολικά στην Ένωση. Η πρότασή μας ε, για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για να υπερασπίσουμε το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών θέλει να συμπληρώσει σημερινή νομοθεσία και για ιδιωτική και για δημόσια επιβολή να καλύψουμε δηλαδή ένα κενό που είχε εντοπιστεί κατόπιν μιας πλήρους ανάλυσης και αξιολόγησης του σημερινού και εκτιμένου για τους καταναλωτές. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε αφενός την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και επαρκή νομική προστασία αφενό για του καταναλωτέ, αλλά αφετέρου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν όλε οι απαραίτητε δικλείδε ασφαλεία για να αποτρέψουμε τι καταχρηστικέ αγωγέ. Επίση, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όσο να τον περισσότερο τη διαδικαστική αυτονομία των κρατών μελών, γιατί αυτό είναι ένα διαδικαστικό μέσο και δεν δημιουργεί ουσιαστικά δικαιώματα για αποζημίωση, απλώς πρόκειται για έναν διαδικαστικό μηχανισμό για συλλογική επιβολή των καταναλωτικών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν έπρεπε όσο δυνατό περισσότερο να διατηρήσουμε το περιθώριο εκτίμησης των κρατών μελών για δικαστικά θέματα και να παρεμβαίνουμε μόνο στις ε, κύριες πτυχές που χρειαζόταν να εναρμονιστούν κατά την άποψή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, Πιστεύουμε ότι έχουμε εδώ μια καλή βάση για συζήτηση για το μέλλον, για τους συνομοθέτες, προκειμένου να τελειοποιήσουμε το νομοθέτημα και επίσης να αποσαφηνίσουμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία. Αν μου επιτρέπετε, στο θέμα της συμπεριλήψης της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των επιβατών στο παράρτημα, γιατί αναφέρθηκε συγκεκριμένα αυτό το θέμα. Όπως ε, βλέπετε, ήδη το επισημάναμε για μελλοντική αξιολόγηση. Όταν αυτό το νομοθέτημα προτείνουμε θα τεθεί σε ισχύ. Γιατί, ε, όπως έχει σήμερα η νομοθεσία, προβλέπει ουσιαστικά δικαιώματα για τους επιβάτες αφενός και κάποιες δυνατότητες απευθεία επιβολή αυτών των δικαιωμάτων σε διμερεί σχέσει μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων αφετέρου. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει δεσμευτικό μηχανισμό και όπω έδειξαν οι εξυλλογήσεις επανειλημμένα, ο τομέας των μεταφορών και των δικαιωμάτων των ευβατών επανειλημμένα παρουσιάζονται ως οι χειρότερες παραβιάσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά δικαιώματα. Επομένως, όντω υπάρχει εδώ ανάγκη για παρέμβαση. Όμως, και πάλι θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις στο μέλλον. Γι' αυτό στην πρόταση το επισημάνουμε αυτό για μελλοντική αξιολόγηση, προκειμένου να αξιολογήσουμε αν υπάρχει συνέπεια, αν υπάρχουν επικαλύψεις και αν χρειάζεται να αναλάβουμε δράση σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής μας έχει το λόγο, ο κύριος Μάγερ. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά όλων σας. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο ακριβώς σε αυτόν τον τομέα να πετύχουμε ισορροπία δυνάμεων και να ε, γίνει αυτό προς όφελος των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην χάνουμε το στόχο μας, τους καταναλωτές δηλαδή. Ε, δεν ε, κατάρτισα την έκθεση, τη γνωμοδότηση μάλλον ε, μόνο. Είναι μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Κυρία Φώστερ, στα σημεία 1, 2, 3 είπα αυτά ακριβώς που είπατε κι εσείς, ότι δεν πρέπει να γίνονται καταχρήσεις των μέσων αυτών, ότι ο καταναλωτής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην συλλογική αυτή αγωγή. Πρέπει δηλαδή να είναι ενημερωμένο, να υπάρχει συγκατάθεσή του. Τέλο, οι εγκεκριμένε οντότητε είπα ότι χρειάζεται να οριστούν. Να, τι ακριβώ ε, καθιστά μια εγκεκριμένη οντότητα και μετά ποιο τη χρηματοδοτεί. Αυτά τα είπα. Μετά, κύριε Βάντεκαμπ, αναφερθήκατε σε ορισμένα θέματα τα οποία, στα οποία θέλω να απαντήσω. Οι αποζημιώσεις αποφασίζονται με, σε στάδια. Πρώτα αποφασίζεται αν κάποιος έχει δικαίωμα αποζημίωσης και μετά καθορίζεται το ύψος της. Τα δικαστήρια είναι αρμόδια γι' αυτό. Μετά, θα προσπαθήσω να ε, συμπεριλάβω τη, τα σχόλιά σας ε, στην έκθεση γνωμοδότηση και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Συγγνώμη κυρία Φώστερ, έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να τα πείτε διμερώς με την Κομισιόν. 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Τροπολογίες για την έκθεση Μέγερ και συνεχίζουμε στην ε, προώθηση της διαφάνειας των ε, επιχειρήσεων, των online επιχειρήσεων υπηρεσιών Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι online πλατφόρμες αποτελούν ένα σημαντικό φορέα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σήμερα, πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τις online πλατφόρμες ως ε, ενδιάμεσος για την υλοποίηση ε, των συναλλαγών. Αυτή η τάση να ε, χρησιμοποιούνται οι online πλατφόρμες μπορεί να οδηγήσει σε μία εξάρτηση των παρόχων υπηρεσιών από τις επιγραμμικές πλατφόρμες για την υλοποίηση των συναλλαγών, κάτι που δημιουργεί ανισορροπία εξουσίας σε ό,τι αφορά τους παράγοντες στην αγορά, έχοντας κατά νου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νομοθετική πράξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προσεγγίζει το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ε, που είναι αντικείμενο online διαμεσολάβησης ε, χρησιμοποιούμε αυτόν τον κανονισμό για να διασφαλίσουμε την ισότητα και τη διαφάνεια για τους παρόχους υπηρεσιών που ε, λειτουργούν μέσω επιγραμμικών πλατφορμών. Ο σημερινός κανονισμός συνεισφέρει στη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ε, ισότητα και την ορθότητα τόσο για τις επιγραμμικές πλατφόρμες όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών. Καταρχήν, θεώρησα απαραίτητο να αποσαφηνίσω και να συμπληρώσω τις ε, διατάξεις ε, μέσω των ε, όρων παροχής υπηρεσιών και μέσω των ιστοσελίδων, έχοντας κατά νου η σημερινή πρόταση, δεν κάνει σαφή διάκριση. Πρότεινα ο όρος του παρόχου μέσω ιστοσελίδας να εκπροσωπεί οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή online επαφή, που σημαίνει οποιαδήποτε software, ιστοσελίδα ή εφαρμογή, ακόμη και στο κινητό, για να προσφερθούν και αγαθά στου καταναλωτέ. Ε, το βρίσκεται αυτό στην τροπολογία 9. Θεώρησε ότι είναι απαραίτητο ο κανονισμό να διασφαλίσει πιο αυξημένο επίπεδο ισότητα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των επιγραμμικών πλατφορμών για, λόγος για τον οποίο θέλησα με την παρούσα έκθεση να τονίσω την ε, ε, αποσαφήνιση κάποιων πτυχών που αφορούν την ισότητα. Και θέλω να αναφέρω και μια άλλη σημαντική πτυχή της έκθεσης, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα διανοητικά δικαιώματα, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. στο brand είναι η καλύτερο ε, τιμή του παρόχου και δεν θα πρέπει να υποχρεούνται οι πάροχοι υπηρεσιών να δίνουν ολόκληρο τον έλεγχο ή μερικό τον έλεγχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε καταγεκριμένα σήματα για να έχουμε αυξημένο επίπεδο ισότητας, θεώρησα καλό να εισάγω μία τροπολογία όπου αναφέρω ότι θα πρέπει οι online πλατφόρμες να ε, χρησιμοποιούν κριτήρια ιεράρχησης των παρόχων υπηρεσιών χωρίς εισαγωγή διακρίσεων. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ιεράρχησης, θα πρέπει να κοινοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών με σαφή τρόπο και εγκαίρος. Για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια σε σχέση με την ιεράρχηση, έχω εισάγει μια τροπολογία η οποία λέει ότι οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση που να προκύπτει από ε, την παροχή λοιπόν πληροφοριών να μην καταλογίζεται στι online σε Ό,τι αφορά τον τουρισμό, θεωρώ ότι η εφαρμογή περιοριστικών κανόνων απέναντι ε, στους παρόχους για την παροχή υπηρεσιών μέσω άλλων διάβλων διανομή, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τη σημερινή αγορά που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό. Κατά την άποψή μου, η ρήτρα του πλέον ευνομούμενου έθνου μειώνει ε, την ανταγωνιστικότητα και περιορίζει την αγορά. Γι' αυτό έχω προτείνει τη διαγραφή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, έχοντα κατά νου σε ορισμένα κράτη-μέλη όπω το Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ήδη υπάρχουν νομοθετικέ προβλέψει στο εθνικό δίκαιο μέσω των οποίων απαγορεύονται ε, τέτοιε ρήτρε. Για την επίτευξη των στόχων τη ψηφιακή ενιαία αγορά. χρειαζόμαστε λύσει ρύθμιση που να είναι εναρμονισμένε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταία πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι η εξή. Επειδή αυτή η πρόταση κανονισμού ε, για να εφαρμαστεί, συγγνώμη, χρειάζονται 12 μήνες, ε, παρά οι 6 μήνες που προτείνονται από την Κομισιόν, καθώς η εφαρμογή μπορεί να σημαίνει πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος. Και Επίσης, ε, επειδή πρέπει να ζητηθεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και να ε, υπάρξει καθορισμός ε, και εκπόνηση νέων εσωτερικών πολιτικών, καθώς και αναθεώρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την προθεσμία εφαρμογής του κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε Κατά τον ίδιο τρόπο έχετε ένα με δύο λεπτά. Κυρία Βιρκούνεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες είναι κάτι πολύ θετικό για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, γιατί τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη αγορά και οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό όμως συνεπάγεται και μεγαλύτερες προκλήσεις. Ορισμένες από αυτές τις επιγραμμικές πλατφόρμες είναι τόσο σημαντικές και μεγάλες που δεν διαπραγματεύονται με τις μικρές επιχειρήσεις. Και οι μεταφορές και ο τουρισμός είναι από τους τομείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από αυτές τις πλατφόρμες. Όταν κάποιος ε, θέλει να ταξιδέψει, κλείνει μόνο του τα εισιτήριά του, το ξενοδοχείο του. Γι' αυτό λοιπόν ε, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το σκηνικό πάρα πολύ. Μετά, οι σχέσεις business to business είναι ε, νομίζω κάτι που ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλύσουν. Ορισμένες πλατφόρμες, όπως είπα, είναι τόσο μεγάλες που δεν διαπραγματεύονται με τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, περισσότερη διαφάνεια, να θεσπιστούν κανόνες. Η Κομισιόν βρίσκεται στο σωστό δρόμο, δεν θέλει να ρυθμίσει τα πάντα, αλλά εστιάζει σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Η σημαντικότερη για μένα είναι οι όροι και προϋποθέσεις. Αυτό το μας το λένε και όλα οι, εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη και η γλώσσα επίσης εύκολη και κατανοητή. Οι όρικοι και προϋποθέσεις επίσης θα πρέπει να κοινοποιούνται στους ε, χρήστες όταν γίνονται αλλαγές ή τροποποιήσεις. Μετά, η βαθμολογίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και χρειάζεται να επέλθει περισσότερη διαφάνεια στον τομέα αυτό. Οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν πώς προκύπτουν αυτές οι βαθμολογίες. Τέλος, πρόσβαση σε δεδομένα. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο δεδομένων και οι χρήστες, οι επιχειρήσεις δηλαδή, δεν τα λαμβάνουν αυτά. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί ποια δεδομένα συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται και από ποιους. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε υπερβολικά στον ε, κλάδο αυτό, όμως ε, πραγματικά χρειάζεται ρύθμιση, διότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ίσος αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Νταμεσμέκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θεωρώ πως η πρόταση είναι καλή αφετηρία για να συνεχίσουμε. Προσωπικά, είμαι υπέρ των, της επιγραμμικής πλατφόρμας και θεωρώ πως είναι μια καλή δυνατότητα για να λύσουμε πολλά, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες βοηθούν τον ανταγωνισμό, βοηθούν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και οι καταναλωτές παίρνουν καλύτερες τιμές. Βέβαια, χρειάζεται να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ε, γίγαντες για να μην ε, καταλήξουμε να μας θυμίζει το σκηνικό τη μάχη Δαβίδη και Γολιάθ. Φυσικά τα κράτη-μέλη έχουν το καθήκον να ρυθμίσουν τον τομέα αυτών με ελάχιστα πρότυπα, έτσι ώστε να καθοριστούν καλύτερα αυτές οι επαγγελματικέ σχέσεις. Η συγγήτρια στη γνωμοδότησή της αναφέρει πολύ σωστά ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η ισορροπία και διαφάνεια στον ανταγωνισμό και χρειάζεται να θεσπιστούν τα ανάλογα μέτρα. Η επαγγελματική χρήση πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Αυτό επίσης είναι σημαντικό και ε, για άλλου τομεί. Πρέπει, α πούμε, να προστατεύσουμε τα εμπορικά μυστικά. Είναι απαραίτητα για την καινοτομία, για τις ε, ιδέες των νεοφυών επιχειρήσεων. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην ενημέρωση των ε, χρηστών, των επαγγελματικών χρηστών. Δεν χρειάζεται υπερβολική ρύθμιση, διότι δεν αποφελείται κανείς από αυτό. Δεν είναι όλοι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μεγάλες εταιρείες γίγαντες. Ε, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο. Για τα υπόλοιπα θα καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και εγώ την δική μας άποψη. Υπάρχει ένα σημείο που θέλω να τονίσω, το οποίο αφορά το σχέδιο της Επιτροπής για... στο σύνολό του. Νομίζω πως πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Δηλαδή έχουμε το eBay απέναντι στον ε, μικρό πάροχο υπηρεσιών. Όμως ε, ας αντιστρέψουμε λίγο την κατάσταση. Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν ορισμένα ιστότοποι μετα-αναζήτησης και είναι πολύ καλή για τους καταναλωτές διότι παρέχουν σύγκριση μεταξύ άλλων ε, ιστοτόπων και ο καταναλωτής καταλήγει να αγοράζει ένα καλύτερο προϊόν σε καλύτερη τιμή υπό καλύτερες συνθήκες. Νομίζω πως ε, αυτή η ιστότοπη μεταναζήτηση ε, ενδεχομένως είναι προβληματική διότι δεν λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες. Όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, υπάρχουν φυσικά και άλλοι τομείς μεταφορών, θα παραμείνω όμως στην αεροπλοεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ειδικέ χρεώσεις, πρόσθετες χρεώσεις από ορισμένε εταιρείε. Και σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον χλιαρά αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Με χαρά μου λοιπόν θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια για να καταφέρουμε να αντιστρέψουμε αυτές ε, τις ε, ισορροπίες προς όφελος των ε, σελίδων αυτών μετα-αναζήτησης, διότι ανταγωνίζονται με αθέμητους όρους τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονιστούν αυτά έτσι ώστε να μην ε, έχουμε στο μυαλό ότι πρόκειται για μεγάλους τεράστιους γίγαντες απέναντι στο μικρό επιχειρηματία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας ανησυχεί κάπως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη θεωρούμε κάπως ήπια. Ιδιαίτερα στον τομέα του, του, τουρισμού και των ε, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και των υπηρεσιών κινητικότητας. υπάρχουν τα πολυτροπικά εισιτήρια, τα οποία επίσης ε, πρέπει να αναφέρουμε, και η αξιολόγηση, η βαθμολογία από αυτές τις ε, πλατφόρμες. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τους εφιστάμενους φορείς τους και να ρυθμίζουν τους τομείς αυτούς ε, εντός των συνόρων τους. Από την άλλη θέλουμε τα τρίτα μέλη να ενημερώνουν τους χρήστες ε, και να μην αφαιρούν το περιεχόμενο από τις ε, πλατφόρμες αυτές αναζήτησης. Πολλές φορές υπάρχουν πολλές κρυμμένες παράμετροι, αλλά εμείς θα θέλαμε να φαίνονται όλα από την αρχή. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμπορικά μυστικά. Αυτά μπορούν να διαγράφονται, να μην φαίνονται αναφερόμαστε στα, στο τελικό προϊόν, το οποίο δεν φαίνεται σε αυτές ε, τις αναζητήσεις. Ορισμένες φορές οι πλατφόρμες ε, έκδοσης εισιτηρίων έχουν κάποια ε, όρια. Εμείς θα θέλαμε να, υπάρχουν, υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός σε αυτά τα όρια. Αναμένουμε λοιπόν τα επόμενα στάδια της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κιλόνεν έχει αποχωρήσει. Θα ήθελα. Ε, κυρία Τσαπαντέλα, θα ε, σας δώσω το λόγο. Μιλάμε για την ψηφιακή επανάσταση και μιλάμε και για ψηφιακές πλατφόρμες. Τι είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα σήμερα. Το πρόβλημα υπάρχει και στον ορισμό. Δηλαδή, ε, αυτό αφορά και την ε, τεχνητή ευφυΐα. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ορισμός. Άρα δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε κάτι που δεν ορίζουμε. Άρα το πρώτο θέμα είναι τι είναι μία ευφυής πλατφόρμα και τι σημαίνει οικονομικό σύστημα που δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλων και μικρών. Άρα υπάρχει η οικονομία της ψηφιακής πλατφόρμας, δηλαδή πολλούμε μία υπηρεσία που δεν είναι μια υπηρεσία μιας ε, της ε, συνεργατικής οικονομίας. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούν την ε, ψηφιακή πλατφόρμα. Το οικονομικό μοντέλο όμως δεν είναι το ίδιο σε σχέση με τη χρήση αυτής της ε, πλατφόρμας. Συνυπάρχουν όμως και γι' αυτό στα οικονομικά πρότυπα ε, δυστυχώς έχουμε το αναδιομένο μοντέλο της συνεργατικής οικονομίας και εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ της μίας και της άλλης, δεν έχει νόημα να ρυθμίσουμε. Υπ' αυτή την έννοια θα υποβάλω τροπολογίες. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο και δίνω το λόγο στον κύριο Κόνιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θίξω τρία σημεία και ευχαριστώ για όλα τα στοιχεία προσκέψη. Πρόκειται για ένα στοχοθετημένο μέσο, δηλαδή η σχέση πλατφόρμας προς επιχείρηση και ζητήματα που ανέκυψαν στην αγορά εργασίας. Δεν πρόκειται για έναν κανονισμό πλατφορμών που θα ορίσει όλα τα θέματα της οικονομίας των πλατφορμών θα υπάρξουν, θα ανακύψουν και άλλες προτάσεις μέσα στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια οριζόντια πρόταση που θα ισχύει για όλους τους τομείς και δεν μιλάμε για ειδικέ λύσεις. Πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι πολύ ελαφρά η προσέγγιση, αλλά είναι το πρώτο σημαντικό βήμα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις επανορθώσεις, που συχνά είναι ένα πρόβλημα για τους χρήστες. Δηλαδή δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους μέσω πλατφορμών και γι' αυτό τα συλλογικά ένδικα μέσα πιέζουν τις πλατφόρμες να βρουν λύσεις. Επίσης δεν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένες απαγορεύσεις και απαγορευτικές ρήτρες γιατί σε αυτή τη δυναμική βιομηχανία δεν θέλαμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ορισμένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν συζητούνται ως προς την ουσία, αν και φυσικά σε ορισμένα κράτη έχουν ληφθεί αποφάσεις. Μία εβδομάδα πριν το παρατηρητήριο για την οικονομία των πλατφορμών ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα ως προς τις διακρίσεις και την πρόσβαση σε δεδομένα καθώς και ρήτρες MFN. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις ανταλλαγές και θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Η κυρία Τσαπαρντέλ έχει το λόγο, τον τελικό λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους, τους κοιόδης. Σημερίζομαι όλες τις προτάσεις που έγιναν όπως σας είπα εξ αρχής και εγώ δεν είμαι υπέρ της υπερβολικής ρύθμισης. Χρειαζόμαστε μια ελάχιστη νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει κατακερματισμός γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη ήδη υπάρχει νομοθεσία που ορίζει αυτές τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης. Χρειαζόμαστε και σαφή ορισμό τι σημαίνει επιγραμμική πλατφόρμα και πώς υπάρχει αυτή η σχέση συνεργασίας μεταξύ πλατφορμών και παρόχων υπηρεσιών. Ε, συνεργαζόμαστε με μικρές σχετικά πλατφόρμες και θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα στα πλαίσια της συνεργατικής ε, οικονομίας. Παράλληλα θα πρέπει να ορίσουμε αυτή τη σχέση συνεργασίας μεταξύ πλατφόρμων και προμηθευτών. Να υπάρχει ε, διαφάνεια και θεμιτός ανταγωνισμός στην ψηφιακή αγορά, δηλαδή μεταξύ ε, παρόχων υπηρεσιών και πλατφορμών. Ο Πάβελ Τέλισκα έφυγε, αλλά θα λάβουμε υπόψη και τα θέματα των πλατφόρμων που συγκρίνουν αγαθά και τιμές όπως υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, αεροπορικά εισιτήρια και ούτω καθεξής. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση και αυτή η ψηφιακή οικονομία θα αναπτύσσεται ένα και περισσότερο. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ ψηφιακής οικονομίας και παλαιών επιχειρηματικών μοντέλων και θα πρέπει να εξεύρουμε τα κατάλληλα μέσα για να εντάξουμε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη νέα ψηφιακή οικονομία που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση θα είναι πολύ καλή προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ταπαρντέλ. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για αυτό το φάκελο είναι στις 17 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε σε ένα σημείο που αφορά την ανταλλαγή απόψεων και θα ζητήσω στους εκπροσώπους της Παγκοσμίας Τράπεζας να έλθουν εδώ στο βήμα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να υποδεκτείτε καταρχήν τον κύριο Ντρες Γκρός, τον κύριο Γκαβίρια και κατόπιν τον κύριο Ελ Χιφνάουι. και τον κύριο Σάιμον Ντέβι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 Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να σας υποδεκτούμε. Όπως ξέρετε η αρχή της συνεργασίας μας είναι από τον Νοεμβρίο του 1997 βάση πρωτοβουλίας ε, του κυρίου Λιμπεράτσκι που είναι εδώ σήμερα. Κύριε Λιμπεράτσκι, σας ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Σήμερα οι συνάδελφοι, γιατί μπορούμε να σας αποκαλούμε συναδέλφους, έτσι. Οι ε, συνάδελφοι λοιπόν από την Παγκοσμία Τράπεζα θα μας παρουσιάσουν τις ε, δραστηριότητες ε, της Παγκοσμία Τράπεζας στον τομέα που μας επασχολεί στον κλάδο των μεταφορών γενικότερα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Ανατολικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να δώσω καταρχήν σε σας το λόγο στον κύριο Γκρός, που είστε διευθυντής του Τμήματος Μεταφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχετε το λόγο και θα είμαι πολύ αυστηρή. Θα χρονομετρήσω γιατί έχουμε ακόμη δουλειά σε αυτή την Επιτροπή. Δέκα λεπτά θα σας δώσω και ε, κατόπιν ίσως μπορούμε να κάνουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους. Θα ήταν τέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια επισκόπηση της δομής ε, της Παγκοσμίας Τράπεζας και της χρηματοδότησης. Ε, έχουμε εδώ τρεις συναδέλφους, τον Χουάνο Γκαβίρια, ο οποίος είναι ε, διευθυντής πρακτικής και η κυρία Κονσάλη είναι Το έχουμε και τους program leaders για την Ανατολική Ευρώπη και τα Ανατολικά Βαλκάνια, τους κυρίους Ελχιφνάφη και Έλλης. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, να ξεκινήσει η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι διεθνές χρηματοοικονομικό ιδρύμα. Έχουμε δύο στόχους, 188 μέλη. Το πρώτο είναι να καταπολεμήσουμε μέχρι το 2030 την ε, απόλυτη φτώχεια και επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί η ευημερία. Θέλουμε λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν ε, υπό ε, πολύ μεγάλες συνθήκες φτώχεια να μειωθούν κατά 2-3%, αλλά θέλουμε επίσης περισσότερη ισότητα έτσι ώστε ε, το κάτω, οι άνθρωποι που είναι στο 40% στο κατώτερο να αυξήσουν το εισόδημά τους. Από το 1994 ιδρυθήκαμε από μια διάσκεψη στο Bretton Woods και τότε μας λέγανε ε, την Διεθνή Τράπεζα για νοικοδόμηση και ανάπτυξη. Η νοικοδόμηση εδώ είναι, είμαστε εδώ, ήμασταν εδώ για να νοικοδομήσουμε Ευρώπη και Ιαπωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ε, να βοηθήσουμε τις λίγες χώρες που είχαν εθνική κυριαρχία, όπως τη Λατινική Αμερική. Ε, μετά, ε, από το 60, επενδύαμε σε εταιρείες με δάνεια που συμμετέχουν σε νοικοδόμηση σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, το 1960, όταν είχαμε την ανεξαρτησία της Αφρικής, ε, προσθέσαμε το AIDA, ε, ουσιαστικά το σκέλος μας soft law που δίνει χρηματοδότηση στις φτωχές χώρες και στο 80 προσθέσαμε την εγγύηση πολυμερών επενδύσεων, προσφέρει εγγύηση σε εταιρείε που θέλουν να επενδύσουν διασυνοριακά και έχουμε ένα κέντρο, το Exit, για τη διευθέτηση της επίλυσης διαφορών. Έχουμε πάρα πολλά γραφεία, πάνω με 100 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ε, τα περισσότερα μέλη μας. Ε, είναι μεγαλύτερος εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, έχουμε την Ιαπωνία στη δεύτερη θέση, την Κίνα στην επόμενη θέση και την Ινδία με 2,3. Οι περισσότεροι μέτοχοι ε, είναι πιο διευρυμένοι. All these lovely black and white photographs you see. Βλέπετε εδώ κάποιες ε, φωτογραφίες ε, από τα project της Παγκόσμια Τράπεζας ε, στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 40 και του 50. Γιατί επικεντρωνόμαστε στις μεταφορές που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη. Καταρχήν προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, μειώνουν την αντιγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς αποδοτικότητα στις μεταφορές. Αλλά αν δούμε πέρα από την Ευρώπη υπάρχει μια τεράστια ατζέντα πρόσβασης. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, κυρίως στην Αφρική, που ζουν χωρίς ε, πρόσβαση σε οδικές ε, μεταφορές και δεν υπάρχει δρόμος. Αλλά ακόμη και εκεί που υπάρχουν ε, υποδομές είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος των μεταφορών. Και δεύτερον, ζούμε ε, στην εποχή της Συμφωνίας Κλίματος των Παρισίων ε, και έχουμε 42 γιγατόνους ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αστρονομικά γρήγορα και την επόμενη δεκαετία αναμένουμε να αυξηθεί κατά 60%. Αν δηλαδή δεν μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα στις μεταφορές δεν θα πετύχουμε τους στόχους των Παρισίων. Φυσικά, το κόστος ε, είναι 1,3 εκατομμύρια. Προκαλεί 1,3 εκατομμύρια νεκρούς ε, ε, στον κόσμο και αυτό ισχύει για τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Ποιοι είναι οι στόχοι μας. Έχουμε τέσσερις στόχους. Καταρχήν, θέλουμε ένα τομέα μεταφορών που να είναι αποτελεσματικό, συμμετοχικό, πράσινο και ασφαλή. Θέλουμε λοιπόν να συνδέσουμε του ανθρώπου με τι αγορέ και τι υπηρεσίε για ε, μεγαλύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο. Εδώ, εμεί ε, είμαστε ο μεγαλύτερο χρηματοδότη. Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 40 δισεκατομμυρίων παγκοσμίω. Πού πάνε αυτά τα χρήματα. Αν πάρετε τα 39 δισεκατομμύρια για να είμαστε ακριβείς, χρηματοδοτούμε περίπου 179 προγράμματα από τα 40 δις, 8,8 δις είναι στην ε, Ανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή και αυτό ε, σε ό,τι αφορά διάφορες ε, υποδομές σε, αστική και μη, σε αστικό και μη αστικό περιβάλλον. Η Ποσαχάρη Αφρική είναι η δεύτερη περιοχή, 8,3 δισεκατομμύρια των επενδύσεών μας. Η μεγαλύτερη περιοχή είναι Κίνα, Κεντρική Ασία και Μογγολία, 7,2 δισεκατομμύρια. 17% των 40 δις, Λατινική Αμερική στη συνέχεια με 5,6 δις και στη Λατινική Αμερική έχουμε περισσότερο αστικές ε, ε, περιοχές, το χάρη ε, χρηματοδοτούμε το μετρό μαζί και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στη συνέχεια έχουμε την Ευρώπη και χώρε κρατημέλη, χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση και τα Δυτικά Βαλκάνια, 3,4 δισεκατομμύρια. Κατόπιν 3 δισεκατομμύρια για την Ασία χωρίς την Κίνα και κατόπιν Αφρική, Πακιστάν περίπου 2,7 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν πέρα από τη χρηματοδότηση θέλουμε να σκεφτούμε ότι και παγκοσμίως αλλά και ευρωπαϊκά συνεισφέρουμε με τις δραστηριότητές μας Έχουμε εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους υποτομείς των μεταφορών. Όταν δανείζουμε λοιπόν στις χώρες ή συνεργαζόμαστε με τι χώρες για την τεχνική βοήθεια ή προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχουμε εμπειρογνωμοσύνη, ε, έχουμε εμπειρογνωμοσύνη σε κάποιους κλάδους όπως είναι η κινητικότητα η αστική. Δηλαδή πώς να έχουμε συστήματα ε, που θα συμπεριλαμβάνει διάφορους τρόπους μεταφοράς και θα αυξήσουμε και τη νέα κινητικότητα σε μια πρόσκοπτη λύση για τους χρήστες. Έχουμε ομάδες εμπειρογνωμοσύνη για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να φτιάξει κανείς ε, μέσα υποδομής, αλλά είναι δύσκολο να τα συντηρήσει. Έχουμε εμπειρογνωμοσύνη ε, για να αναπτύξουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση. Έτσι λοιπόν, πώς θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε οικονομικά ωφέλη ε, στην πόλη. Επίση, έχουμε ειδικού για την οδική ασφάλεια. Μου άρεσε η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή πριν να ξεκινήσουμε για την οδική ασφάλεια. Είναι τεράστιο θέμα παγκοσμίω, 1,3 εκατομμύρια θύματα παγκοσμίω και έχουμε και ειδικού στην πράσινη μεταφορά, στις πράσινες μεταφορές. Δεν δείτε τώρα δεξιά στην οθόνη τις κοινότητα πρακτική. Εδώ έχουμε άλλου τομεί το φύλλο. Ποιο φύλλο θα μου πείτε. Ουσιαστικά θέλουμε οι μεταφορές να συμπεριλαμβάνουν και τα δύο φύλλα. Δηλαδή έχουμε παραδείγματο χάρη υπόγειες διαβάσεις, αλλά πώς θα χρησιμοποιήσουν τις διαβάσεις οι γυναίκες και δεν αισθάνονται ασφαλής. Επίσης, ε, επίλυση σειράξεων, αντιμετώπιση της βίας, ε, κυρίως στο Κογκό, στην ε, Αφρική ή σε περιοχές που δραστηριοποιείται η Μπόκο Χάραμ στο Καμερούν. Ε, παραδείγματο χάρη θα πρέπει να ε, δεις ε, πώς θα αντιμετωπίσει τις απαγωγές. Επίσης έχουμε ειδικού στην μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στην Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης η ανάπτυξη που προσανατολίζεται στο τράνσιτ. Μπορείς να έχεις διάφορους διαδρόμους, αλλά πώς θα έχεις αστική ανάπτυξη που να λειτουργεί βάσει της ραχοκοκαλιάς των υποδομών. Και τέλο, έχουμε ειδικού στη διαχείριση των συμβάσεων Πώ πώς ε, να έχουμε τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες ε, σε μεγάλα έργα υποδομής. Και νομίζω ότι είναι αυτή η τελευταία διαφάνεια για την επισκόπηση. Έτσι λοιπόν, ε, σας εξοικονόμησα και ένα μισή λεπτό, θα το δώσω στο συνάδελφο. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής Μεταφορών θα σας μιλήσω για τις επενδύσεις ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, αποκλίνουσες τάσεις που διαγράφουν. Από το 49 και μετά, 47 και μετά, με συγχωρείτε, η Παγκόσμια Τράπεζα είχε μακροχρόνιες δεσμεύσεις ε, στα τότε κράτη-μέλη. Στη συνέχεια είχαμε και άλλες προσχωρήσεις και φυσικά θέλουμε να δούμε τα ε, παγκόσμια, τις παγκόσμιες τάσεις ζήτησης ε, ανάλογα με τα ιδρυτικά μέλη ή τα κράτη τα οποία προσχώρησαν στη συνέχεια στις επόμενες δεκαετίες. Όπως βλέπετε τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πολύ λιγότερα από τις προηγούμενες ε, δεκαετίες. Ποιος είναι ο ρόλος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι αναδιόμενες ε, τάσεις. Καταρχήν θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις ε, καθολικές γνώσεις μέσα στα πλαίσια των ε, αναπτυξιακών λύσεων. Πολλά, μέσα σε πολλά προγράμματα θέλουμε να υποστηρίξουμε τις πολυσχηδείς διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, ε, να καλύψουμε τα επενδυτικά κενά, ιδιαίτερα στις ε, περιοχές που έχουν μείνει πίσω και την ενίσχυση των θεσμικών πλαισίων, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που προσχώρησαν πιο πρόσφατα Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία και επίσης να μάθουμε από την Ευρώπη και να προσαρμοστούμε στα πλαίσια χαμηλότερων εισοδημάτων, δηλαδή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα για να αναπτυχθούν λύσεις για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Την τελευταία δεκαετία στο λιμάνι της Ριέκα, στην ε, Κροατία, έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα. Τι κάνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία σειρά ε, προγραμματών γνώσεων, δηλαδή τεχνική αρρωγή και χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη μέσω ε, διαχείρισης της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας για την οδική ασφάλεια, για την ε, διαχείριση ατυχημάτων και ούτω καθεξής. Επίσης έχουμε 8 με 10 επιχειρησιακά προγράμματα. Φέτος είχαμε μόνο ένα και έχουμε και διάφορες δραστηριότητες, ε, ενεργά προγράμματα και έχουμε και ASAs, ε, δηλαδή αναλυτικές, αναλυτικά προγράμματα υποστήριξης στις χώρες γειτονίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 2,8 ε, δις μέσα στα πλαίσια των επίγειων μεταφορών και των ε, ε, διάβλων, οδικών μεταφορών, σιδηροδρομικών και ούτω καθεξής. Αυτό αφορά και τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, όπως την Κροατία που σας προανέφερα, και τεχνική αρρωγή ή ε, πολυτομιακές παρεμβάσεις. Άρα ποια είναι τα αναδυόμενα θέματα. Καταρχήν, όπως είπατε και νωρίτερα, στην Επιτροπή Μεταφορών είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, ακόμα και σε προηγμένο περιβάλλον. Πολλές φορές ε, ζητάμε λύσεις σε πιο ενισχυμένα πλαίσια, σχηδή πλαίσια. δηλαδή τη μεταρρύθμιση μεγάλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ως προς τις κοινωνικές υποχρεώσεις, θέματα εξυγχρονισμού μεταφορών, ψηφιακές πλατφόρμες για την οδική ασφάλεια, υποδομές, ενδεικτικά σχέδια και ούτω καθεξής. Ε, δηλαδή υπάρχουν συνεκτικά προγράμματα, αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και να εφαρμόσουμε άμεσα αυτή την καθολική γνώση. Πρόκειται για δύσκολα προγράμματα και θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή να μιλάμε με μία φωνή έτσι ώστε να εισακουστούμε καλύτερα. Επίσης, οι εταιρικέ σχέσεις και υποστήριξη οδηγούν σε καλύτερη χρηματοδότηση. Έχουμε δηλαδή κοινή ε, χρηματοδότηση με την ε, Τράπεζα Ανάπτυξης και με άλλους θεσμούς και μπορούμε να έχουμε και συμπληρωματικά ε, μέσα χρηματοδότησης που έχουν μεγάλη σημασία για να καθορίσουμε την τάση αυτή. Υπάρχουν ε, βέβαια και συμπληρωματικές δεξιότητες, για παράδειγμα ασχολούμαστε με την ε, ε, συρρήκνωση που υπάρχει στα εργασιακά και γι' αυτό χρειάζονται συμπληρωματικές δεξιότητες σε ρυθμιστικά πλαίσια. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να έχουν αποκλίνουσες απόψεις ή άλλες προτεραιότητες Υπάρχει το πλεονέκτημα να μαθαίνουμε ημέν από τους δε, να προωθήσουμε την καινοτομία μέσω από διαφορετικές θεωρήσεις και επίσης, ε, ας πούμε, στον ψηφιακό κόσμο και τις μεταφορές, το 2018 υπάρχουν νέες εξελίξεις. Άρα, η η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να προωθήσει θέματα πέρα από τη χρηματοδότηση της τάξης των ε, επιδοτήσεων, των ε, κοινοτικών επιδοτήσεων. Με τη Βουλγαρία ασχολούμαστε με το θέμα της ε, ηλεκτρονικής, των ηλεκτρονικών διοδίων, έτσι ώστε να ανοίξουμε νέες διόδους και νέες δυνατότητες. Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις. Φυσικά Ω ως προς τις πράσινες μεταφορές, ο τομέας αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθούμε τα αναπτυξιακά πρότυπα και να χρηματοδοτήσουμε νέες λύσεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργαζόμαστε σε επιμελητιακά ζητήματα, δηλαδή τον διάδρομο TEN-T, για να δώσουμε κίνητρα και ε, να κάνουμε μία ιεράρχηση των επενδυτικών σχεδίων και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την ποιότητα τη ζωή των πολιτών, κινητικότητα και διαχωρισμό των φύλων, έτσι ώστε να εισαγάγουμε και το στοιχείο αυτό του φύλου και μας απασχολεί και η περιφερειακή ολοκλήρωση και οι περιοχές που έχουν μείνει πίσω, οδική ασφάλεια και μεταρρυθμίσεις στον σιδηροδρομικό τομέα, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, πιο πράσινη ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να συνεργαστούμε με τις ε, χώρες που έχουν μείνει πίσω στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ δεν ξεπέρασα το χρόνο μου. Ο κύριος Έλλης για οικονομία χρόνου θα κάνει μόνο του την παρουσίαση και θα χρησιμοποιήσει και τα 10 λεπτά που έχει στη διάθεσή του. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ναι, ναι, να σας υπενθυμίσω ότι όταν είπα 10 λεπτά εννοούσα μια γενική παρουσίαση Πρέπει να έχουμε το χρόνο για να συζητήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν κάντε τα 10 λεπτά 5. Πώς το βρίσκετε. Καλή συμφωνία. Okay, I'm, um, I'm Θα τα πω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας μιλήσω για τις, ε, τη τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Επόμενη διαφάνεια. Ε, Πώ δραστηριοποιούμαστε στι χώρε αυτέ. Διαφέρει λίγο η δράση μα από την δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι διαφέρουν οι υποδομές, τα κενά από αυτόν, η πολιτική ε, και οι συνθήκε. Γι' αυτό λοιπόν ε, υπάρχουν ιδιαιτερότητε, τι οποίε δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αν δεν συνεργαστούμε με τι κυβερνήσει. Συνεργαζόμαστε με τι κυβερνήσει ή του πελάτε μα, δηλαδή, τη Γενική Διεύθυνση NIR, τη Γενική Διεύθυνση MOVE, δίκτυα μεταφορών που στηρίζουν την ε, ιεράρχηση των ε, προτεραιοτήτων στις ε, μεταφορές στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει το παρατηρητήριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το πάνελ για τις μεταφορές στις περιοχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι φορείς συμμετέχουν στις δράσεις μας. Κύρια χαρακτηριστικά των χωρών αυτών είναι η μεγάλη αποκέντρωση που λαμβάνει η χώρα τελευταία. Υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες που περνάνε από το εθνικό το τοπικό επίπεδο, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες ε, και υποδομές γι' αυτό. Η Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθεί να φέρει κοντά τους σε διάφορους εταίρους. Για παράδειγμα, στη Σερβία πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα συνέδριο με τίτλο «Κατανοώντας τον κίνδυνο» όπου συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες και τα ευάλωτα σημεία των Δυτικών Βαλκανίων. Ενδεικτικά αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά το δανεισμό, ε, δανείζουμε και για συγκεκριμένα έργα αλλά και για προγράμματα. Υπάρχει εστίαση πολιτικής, υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και φυσικά ε, οι αναλύσεις που διεξάγουμε, οι οποίες είναι πολλές. Επόμενη διαφάνεια. Πολύ σύντομα. Η συνδεσιμότητα σε περιφερειακό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τις χώρες αυτές με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται πολλά για την ε, διαχείριση των συνόρων, ε, μεθοριακούς ελέγχους, βελτίωση των υποδομών. Ε, συντήρηση του οδικού δικτύου, πολλές επενδύσεις ε, προορίζονται για τη δημιουργία νέων διαδρόμων, αλλά υποχρηματοδοτείται η συντήρηση των υποδομών αυτών. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε αυτό. Αν έχετε ταξιδέψει στα Δυτικά Βαλκάνια θα, ε, καταλάβετε ότι η ανθεκτικότητα και η, στο, στις καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι από τις πιο ε, είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη μόλυνση στην Ευρώπη, οπότε προσπαθούμε μέσω επενδύσεων για τη βελτίωση, για παράδειγμα, των δημόσιων συγκοινωνιών, να αλλάξουμε την κατάσταση. Εδώ βλέπετε ένα κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βοσνία και δεν ξέρω αν το πιστεύετε ή όχι. Αυτό είναι σταθμός, αυτή είναι η αποβάθρα που βλέπετε. Προσπαθούμε λοιπόν να αλλάξουμε την ε, ταχύ επιδείνωση των συνθήκων και των υποδομών στα Δυτικά Βαλκάνια. Μετά, μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων. Το θέμα δεν είναι μόνο η συντήρηση του δικτύου ή η δημιουργία καινούργιου, αλλά και η μεταρρύθμιση των ε, επιχειρήσεων των ε, σιδηροδρόμων. Μετά, προσπαθούμε να επιτύχουμε συνδεσιμότητα σε τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούμε με τους Δήμους και τις κοινότητες για να στηρίξουμε τον τουρισμό, τη γεωργία και την εκπαίδευση και ε, να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις μας θα ε, έχουν υπόψη τους και αυτούς τους τομείς. Μετά, στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας δραστηριοποιούμαστε αρκετά τον τελευταίο καιρό. Συνεργαζόμαστε με την DigiMove και την DigiRegio για προγράμματα τα οποία, τα οποία περιλαμβάνουν ιεράρχηση και αξιολόγηση των στόχων. Θέλουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας και γι' αυτό προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τη συμμετοχή όλων των ε, σημαντικών φορέων και εταίρων στις περιοχές αυτές. Μετά, οδική ασφάλεια, πολύ σημαντικό τομέας των δραστηριοτήτων μας τα θύματα από τροχέα στις χώρες αυτές είναι δύο και τρεις φορές περισσότερα από ό,τι σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρονται προβλήματα στην επιβολή του νόμου. Συζητάμε το ενδεχόμενο αυτόματης επιβολής ορίου ταχύτητας έτσι ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από Φυσικά ε, φροντίζουμε και στον τομέα της τεχνολογίας να έχουμε πρόσβαση στα μαύρα κουτιά. Μετά, ε, φοδιαστική, δίνουμε έμφαση σε αυτό. Ορισμένες χώρες έχουν σημαντικές ελλείψεις και αυτό φαίνεται στα συστήματα μεταφορών. Επόμενη διαφάνεια. Και άλλη. Πιο πέρα. Τουρκία. Τελευταία διαφάνεια. Είναι η Σμύρνη το μέρος που βλέπετε εδώ είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε για ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό και ΕΦΗ συστήματα μεταφορών. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές, την αρχιτεκτονική των συστημάτων στο δικό δίκτυο και τους σιδηροδρόμους. Νομίζω πως δεν έχω άλλο χρόνο, γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Χρήζεται χειροκροτή Και αφήσω και στον συνάδελφό σας πέντε λεπτά για να πάρει το λόγο. Α, δεν θέλετε. Μάλιστα, πολύ σπάνιο να αρνείστε το χρόνο αγόρευση από την πλευρά τη Παγκοσμία Τράπεζας. Λοιπόν, θα περάσουμε στη συζήτηση με τα μέλη τη επιτροπή. Ο κύριος Βαντεκάμπ, ξεκινήστε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, τα θερμότατα συγχαρητήριά μου στον κύριο Λιμπεράτσκι, ο οποίος είναι υπεύθυνο και διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης. Νομίζω πως ε, οι παρουσιάσεις από τους τέσσερις προσκεκλημένους είναι εντυπωσιακότατες. Δυστυχώς δεν επιτύχαμε ισότητα και τέσσερις άντρες είναι, αλλά ας το προσπεράσουμε. Να σας πω ότι όταν ήμουν στο γυμνάσιο άκουσα για τη συμφωνία του Bretton Woods που θα βοηθούσε τις πιο αδύναμες περιοχές. Γι' αυτό προς τους ε, εκπροσώπους της Παγκόσμια Τράπεζας. Δεν έχω καταλάβει τι κάνετε ακριβώς εντό ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πω ε, παρά είμαστε πλούσιοι και αν θέλετε τεμπέληδε για εσά, μήπως θα έπρεπε να δώσετε έμφαση σε άλλες χώρες όπως το Μπαγκλαντέ η Μιανμάρ, χώρε της Αφρικής. Τι κάνετε εδώ στην πλούσια Δύση η Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ουκρανία είναι χώρε που μπορώ να κατανοήσω γιατί δραστηριοποιείστε. Όμω εντό Ευρωπαϊκή Ένωση τι ακριβώ κάνετε. Έπικα. Είχαμε εκπροσώπους της ΕΤΕΠ εδώ και αγχώνομαι πάντα όταν συνειδητοποιώ ότι η ΕΤΕΠ έχει και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε κέρδος από όλες αυτές τις επενδύσεις. Τρίτη ερώτηση, πώς είναι η συνεργασία με την ΕΤΕΠ, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας, διότι καταλαβαίνω πως η Παγκόσμια Τράπεζα έχει άλλες προτεραιότητες ε, χρηματοδότησης από την ΕΤΕΠ και άλλα κονδύλια. Τέλος, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας που πήγε στην Κίνα και εκεί ήρθαμε αντιμέτωποι με, την ε, Ασία, με τις ασιατικές υποδομές και την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Πώς είναι η συνεργασία σας με την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι ένα ίδρυμα κομμουνιστικής χώρας ε, και κατηγορείται ότι προσπαθεί να ε, εισβάλλει απεικιοκρατικά στην Ευρώπη. Η κυρία Λουκατσάνσκα. Ευχαριστούμε κύριε Βαντεκά, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η Παγκοσμία Τράπεζα κάνει πολλά και έχει κάνει πολλά και για τη δική μου περιφέρεια πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνατε πολλά για τις υποδομές στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και τώρα έχουμε τέσσερις χώρες, Βουλγαρία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία, που εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα δικά σας κονδύλια. Στην ιστοσελίδα σας βρήκα κάποιες πληροφορίες ε, για τη χώρα μου, την Πολωνία. Διάβασα ότι το τελευταίο project για τις μεταφορές εφαρμόστηκε το 2015. Είχε υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχει κάποια δραστηριότητα που να λαμβάνει τώρα χώρα σε αυτή την ε, περιοχή. Η σημερινή κυβέρνηση είναι ενεργή στον τομέα. Προσπαθούν να χτυπήσουν την πόρτα σας να ζητήσουν χρηματοδότηση για project για έργα μεταφορών ή καθόλου. Και δεύτερη ερώτηση. Συναντάστε με άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάτε για την αναγκαιότητα να καταπολεμήσετε την ατμοσφαιρική ρήπανση, τον έφος. Υπάρχει κάποιο δικό μέσο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκηση, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Υπάρχει ένα τέτοιο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση τη ατμοσφαιρική ρήπανση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ήθελα να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά τι γίνεται με το αν υπάρχει μια ε, ολοκλήρωση σε σχέση με τα κονδύλια που έχουν να κάνουν με την προσχώρηση. Και επίσης μια ερώτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να καταλάβω ποιο σύνδεσμο υπάρχει με τι κινέζικε επενδύσει. Παραδείγματο χάρη για την ε, οδό του μεταξιού. Γιατί σίγουρα προτιμούν τη θαλάσσια εδώ, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η Κίνα χρησιμοποιεί και εναλλακτικέ οδού, δηλαδή επενδύσει ε, χερσαίε. Επομένως, ε, τι γιατί επενδύσεις κυρίως μιλάμε, πρόκειται για άμεσες επενδύσεις ή για χρηματοδοτήσεις και θα ήθελα και την άποψή σας ε, σε ό,τι αφορά την κοινότητα μεταφορών που δημιουργήθηκε μετά τη διαδικασία του Βερολίνου για να καταλάβω αν αυτή η κοινότητα, αυτός ο νέος οργανισμός είναι ενεργός. Έχετε σχέσεις με αυτούς. Και επίση, ποιε είναι οι εσωτερικές σχέσει με τα Δυτικά Βαλκάνια. Θυμάμαι μια ωραία διακοινοβουλευτική διάσκεψη που έλαβε χώρα στην ε, Πρίστινα και είναι κάτι ε, που μας ε, έχει απασχολήσει εμάς ως Επίμετρα και ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση στο ποιος επενδύει περισσότερο στους σιδηροδρόμους ή περισσότερο σε οδικές μεταφορές και πώς ε, αλλάζουν οι επενδύσεις ε, αν κάποια χώρα πλησιάζει περισσότερο ή λιγότερο ε, στην ένταξη. Είδαμε και τι έγινε με το δημοψήφισμα στις 30 Σεπτεμβρίου στη Φύρομ. Τι αλλάζει για σας και μια ερώτηση για τον τουρισμό. Τι είδους επενδύσεις υλοποιείτε και τι είδους ε, επιρροή ε, απαντάτε. Δηλαδή, στο Μαυροβούνιο έχουμε χώρες, από, έχουμε συγγνώμη, επενδύσεις από τις χώρες του κόλπου. Ε, ε Παραδείγματο χάρη γίνεται μια επένδυση για τη σύνδεση, αλλά είχαμε και μια τουριστική επένδυση. Θα ήθελα λοιπόν την αξιολογησή σας και για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ντεμόντε. Κύριος Κίστιλορ. Yes, of course. Thank you very much, Chair, Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Βλέπω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθεί να φτάσει στην ισότητα των φύλων στο μέα των ε, μεταφόρων. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έγινε και στη δική σας οργάνωση, γιατί βλέπω ότι στην αντιπροσωπεία σας είσαστε μόνο άντρες. Αυτό είναι αποδεκτό. Έχετε γυναίκες συναδέλφους και αν ε, όχι, γιατί όχι γιατί δεν είναι εδώ. Αυτά. Bon, ça ε, επειδή όμως ε, γυναίκα προεδρεύει την Επιτροπή σας, να, ε, διαφοροποιείται το πάνελ εδώ, τα έδρανα εδώ. Κύριε Βαντεκάμπ, τι θέλετε να μου πείτε. Κύριε Λιμπεράτσκι, θα μας ε, πείτε και εσείς λίγα λόγια, γιατί είναι δική σας η καλεσμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή εισαγωγική σας ε, παρατήρηση. Η κυρία Κάρλα Γκονσάλες Κάρλα Χάλτ είναι και αυτή ε, παρούσα, άρα δεν είναι μόνο άντρες ε, παρόντες από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ευχαριστώ και τον κύριο Βαντεκάμπ. Γιατί είναι εδώ η Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμιας Τράπεζας και Ήθελα να έχουμε μακροχρόνιες επαφές με την Παγκόσμια Τράπεζα. Γιατί πρώτη, οι πρώτες μεταφορές, μα αυτό είναι αυταπόδεικτο. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και ειδικά ένα. Στην ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης μου θα ήθελα να πω ακριβώς τα ίδια λόγια. Έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες ασφαλείς μεταφορές, πράσινες μεταφορές, μεταφορές ε, ε, γενικότερα και όπως καταλαβαίνετε η Παγκόσμια Τράπεζα επιθυμεί να ευεργετεί. Είναι ευεργετών ε, ο οργανισμός και όχι κερδοσκοπικός. Μας ενδιαφέρουν οι διάβλοι μεταφοράς, τι αφορά την Ευρώπη, η διάβλη μεταφορών και οι σχέσεις με τη γειτονία, όπως παρουσιάσετε εδώ μέσα στα πλαίσια συνεκτικών δικτύων, δηλαδή ε, τις διατροπικές μεταφορές σιδηροδρομικές ε, εσωτερικών πλωτών οδών, θαλασσίων και ούτω καθεξής. Εσείς θέλετε να μάθετε και από την ευρωπαϊκή πείρα, επειδή υπάρχει, υπάρχει πείρα από δικής μας πλευράς ε, σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, τις διατροπικές μεταφορές, θαλάσσιες, πλωτές και ούτω καθεξής. Έχουμε πολλά κοινά μεταφορά αγαθών κυρίως και φυσικά μιλάμε για λογικές τιμές έτσι ώστε να φτάσουμε σε ευημερία και σε κέρδη για να έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλα τα μέλη που έλαβαν το λόγο. Ε, κυρία και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δώσατε να, συμμετάσχετε, να συμμετάσχουμε όλοι εδώ σε αυτή τη συζήτηση και στις 6.30 προβλέπεται δεξίωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιμπαράτσκι. Και η πρόεδρος έχει μία ερώτηση. Μιλήσατε για τους στόχους σας προς επίτευξη, αλλά πώς επιλέγετε τα προγράμματα, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής Υπάρχει η κλιματική πρόκληση, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Μιλήσατε για βιώσιμο σχέδιο αστικών μεταφορών. Σας ασχόλησαν και οι αγροτικές μεταφορές που είναι πρόκληση του 21ου αιώνα. Και ποιες είναι οι προπτικές. Ε, κάνετε προβολές προς το μέλλον σε 10-20 χρόνια το αυτοκίνητο δεν θα υπάρχει πλέον. Θα έχουμε αυτόνομη οδήγηση, θα έχουμε μια άλλη μορφή κινητικότητας. Αυτά τα σενάρια τα λαμβάνετε υπόψη για να προσανατολίσετε κυβερνήσεις που σας προτείνουν παλαιά σχέδια 40 ετών πριν για τις οδικές μεταφορές, τις αεροπορικές. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη διακυβέρνηση σε περιφερειακό επίπεδο ή κρατικό. Δηλαδή τέσσερις είναι ερωτήσεις και όχι μία. Ποιος θα αρχίσει. Θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα περάσω στους συναδέλφους να πατήσουν εκείνη τα δύσκολα. Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στη δική σας ερώτηση πρώτα. Πώς επιλέγουμε τα project που χρηματοδοτούμε. 189 μέλη έχει η Παγκόσμια Τράπεζα, 120 χώρες είναι εκεί όπου τρέχουν διάφορα και υπάρχει και ένα πλαίσιο. Ε, υπάρχει ένας χρηματοδοτικός φάκελος ε, που διαθέτουμε για την κάθε χώρα, οπότε τους ρωτάμε πώς θέλετε το χρησιμοποιήσουμε. Ε, είναι οι προτεραιότητε τη κάθε χώρα, πλούσια, φτωχή ή κάπου στη μέση. Ο τομέας των μεταφορών, ας πούμε, είναι ένας τομέας όπου η έμφαση είναι στο πρασίνισμα, σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον, μεταφορές, σε μείωση των εκπομπών. Επίσης, έχουμε διαμορφώσει ένα συνασπισμό πριν από μερικούς μήνες, στον οποίο συμμετέχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επενδυτικές τράπεζες από όλο τον κόσμο και το λέμε Zoom for All, βιωσιμότητα και κινητικότητα για όλους. Προσπαθούμε να εστιάσουμε και στο περιβάλλον, στο πρασίνισμα, στην προσβασιμότητα, στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε αυτούς τους τέσσερις τομείς. Κοιτάζουμε τις επιδόσεις κάθε χώρα σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, τέσσερις τομείς και καταρτίζουμε σχέδια δράσης για τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα βασικά, ε, βασικές ανάγκες της κάθε χώρας και ε, αρχίζουμε το σχεδιασμό από εκεί. Αυτά έτσι γενικότερα. Κύριε Λιμπεράτσκι, ρωτήσατε γιατί μας αρέσει να δουλεύουμε στην Ευρώπη. Γιατί ε, είναι ένα σημαντικό εταίρος, είναι μια προχωρημένη περιοχή και μπορούμε να μάθουμε πολλά από εσάς και να μεταδώσουμε τις γνώσεις αυτές σε άλλες χώρες. Ένα παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες, ήμου, μάλλον πήγα για δύο εβδομάδες στον Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα και άντλησα από την πρόσφατη εμπειρία μου στην Κροατία όπου επαναχρηματοδοτήθηκε χρέος από ε, επιχειρήσεις που είχαν κηρύξει πτώχευση μέσω ενός πολύ έφιου συστήματος. Η Παγκόσμια Τράπεζα επέτρεψε την επαναχρηματοδότηση αυτών των εταιριών. Και κατάφερε να μοχλεύσει την αγορά έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Αυτή είναι πολύ συναρπαστικά. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μεταφέρουμε τη γνώση αυτή και στις άλλες χώρες. Για παράδειγμα στη Σρι Λάγκα και στην ε, Ινδονησία που πήγα. Τώρα, δεν γνωρίζω την ακριβή θέση τη ΕΤΕΠ για τη χρηματοδότηση, όμω είπα στην Παγκόσμια Τράπεζα τα πράγματα έχουν ω εξή. Όλα τα μέλη μα και οι 28 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συνεισφέρει 17 δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό μας. Τα 7,5 θα πληρωθούν σε βάθος χρόνου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με 17 δις κεφάλαιο, τα οποία καταβάλλονται από το 1944 και μετά. Έχουμε κερδίσει χρήματα από δάνεια που δώσαμε σε πιο πλούσιες χώρες. Τα επαναδιοχετεύσαμε ε, στο κεφάλαιό μας και ε, σε αυτό προστίθενται και τα κέρδη από τις επιχειρήσεις μας. Μετά, όταν δανείζουμε σε χώρες με υψηλό εισόδημα, χρησιμοποιούμε τη διαφορά και χρηματοδοτούμε τις φτωχότερες. Από τα κέρδη δηλαδή του δανεισμού ε, προς το Μεξικό, προς την Κίνα, προς τις χώρες δωρητές που έχουν δηλαδή συνεισφέρει στο ε, κεφάλαιο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα χρήματα λοιπόν που διοχετεύτηκαν στη, στο EBRD είναι λιγότερα από τα χρήματα που επενδύθηκαν στις ε, χώρες που το είχαν ανάγκη. Τώρα, κύριε Βάντεκαμπ, ε, στο γυμνάσιο μάθατε πως είμαστε η τράπεζα των φτωχών. Ναι, επενδύσαμε 25 δις δολάρια σε χώρες όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μετά, δραστηριοποιηθήκαμε και σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα. Αλλά όταν κάποιος, ας πούμε, μια πλούσια χώρα έχει πρόσβαση σε ενταξιακά κονδύλια, δεν θα έρθει σε εμά. Θα πάει σε εμά ε, όχι επειδή έχει έτσι μια μικρή δυσκολία. Θα, θα έρθουν σε εμά επειδή έχουν μεγάλα προβλήματα και θέλουν βοήθεια και τεχνική υποστήριξη. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται χώρες σε εμά. Μέχρι και η Κίνα θέλει να δανειστεί από εμά. 1,5 δι δανείστηκε πρόσφατα ε, και μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να μας αγοράσει και να αγοράσει 10 τράπεζες σαν και εμά. Όμως δανείζονται από εμά γιατί θέλουν να δουν πώς μπορούν να ε, ενσωματώσουν στον ε, σχεδιασμό τους διάφορους τρόπους μεταφορών και την τεχνογνωσία αυτή μετά μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ε, σε άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ΕΤΕΠ, όπως γνωρίζετε, μόνο γύρω στα δύο χρόνια λειτουργεί. Υπάρχει κεφάλαιο, αλλά τα πρότυπά τους είναι υψηλά. Δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Νομίζω τελευταία φορά που το ψάξα ήταν περίπου 200 υπάλληλοι στην ΕΤΕΠ. Τα project λοιπόν που χρηματοδοτεί είναι, είναι επιλεγμένα. Μέχρι τώρα δεν έχει επενδυθεί τίποτα ε, σε ορισμένους τομείς. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ασίας, εμείς και κάποιες ε, λίγες άλλες τράπεζες ε, έχουμε αναλάβει τον όγκο της χρηματοδότησης. Με την ΕΤΕΠ συνεργαζόμαστε στενά. Ήμουν υπεύθυνο τη ε, Παγκόσμια Τράπεζα για τα νησιά του Ειρηνικού, Παππού, Νέα Γουινέα κτλ. Και ε, εκεί χρηματοδοτούμε έργα υποδομής, αλλά και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, α πούμε, στο Εκουαδόρ χρηματοδοτούμε ε, σχέδια υπόγειου σιδηρόδρομου, σχέδια δημόσιων συγκοινωνιών και νομίζω πως μπορούμε να βρούμε στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνουν και τους ε, δυο μας. Τώρα, ε, έγινε μια ερώτηση για την Πολωνία και άλλη μια για την ενσωμάτωση των ε, κονδυλίων. Θα δώσω όμως το λόγο στους ε, συναδέλφους μου για να τις απαντήσουν. Λοιπόν, ε, για την ερώτηση της ε, κυρίας από την Πολωνία. Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί πριν λίγο καιρό συμμετείχαμε σε ένα μεγάλο έργο αναδιάρθρωσης των σιδηροδρόμων. Αυτό ήταν ε, ίσως ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα αναδιάρθρωσης σιδηροδρόμων που υλοποιήσαμε και επιτυχώς γιατί νομίζω ότι ε, ήταν ε, η εταιρεία τότε δεσμευμένη στις, υποχρεω... στις κοινωνικές δεσμεύσεις και εμείς ε, παρακολουθήσαμε και συνοδεύσαμε αυτό το έργο και είχαμε και ένα άλλο έργο ε, για τους δρόμους και για την ερώτησή σας τι κάνουμε από τότε. Όπως ε, ξέρετε, λόγω του χαμηλού εισοδήματος στην Πολωνία εργαστήκαμε κυρίως σε περιοχές πιο φτωχές και υλοποιήσαμε ένα σχέδιο τεχνικής βοήθειας που καλύπτει τέσσερις πόλεις στην Πολωνία Συγγνώμη για την προφορά μου, το Μπάλιστοκ, Λούμπλιν, Σέσο και Όλσιν, τις πόλεις αυτές. Και ουσιαστικά εξετάσαμε τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας και προτείναμε κάποια, ε, κάποιες τροποποιήσεις και πιο πρόσφατα με την πολωνική κυβέρνηση κάναμε μια ανάλυση για να ενισχύσουμε ένα πρόγραμμα που αφορά τις χερσαίες οδούς. Ε, είχε να κάνει και στη συνεργασία με, Ευρωπαϊκή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Εθνικές Οδούς στην Πολωνία. Και προτείναμε στην κυβέρνηση ένα τέτοιο πρόγραμμα για να δούμε αν ενδιαφέρονται να έχουν και την υποστήριξη της Παγκοσμίας Τράπεζας. Αυτά που ρώτησε η κυρία Ντεμοντέ για το Μαυροβούνιο. Στην περίπτωση των μεταφορών συγκεκριμένα δεν συμμετέχουμε, όμως πρέπει να πω ότι στην περίπτωση του Μαυροβουνίου αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο έργο μεταφορών που χρηματοδοτείται από άλλες πηγές χρηματοδότησης και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην δημοσιονομική θέση της χώρας και εξαιτία αυτού δεν συμμετέχουμε εμείς στον κλάδο των μεταφορών. Όμω είμαστε πολύ ενεργοί σε άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων στον τομέα των μεταφορών. Ξέχασα να απαντήσω στον κύριο Τέιλορ για το θέμα του φίλου. Είναι ντροπιαστικό αυτό το πάνελ, τέσσερις άντρες με σκούρα κουστούμια. Αλλά να πω από τους ε, δέκα διευθυντές μας ε, της Global Practice, οι τρεις ε, είναι γυναίκες. Ε, θα έπρεπε να έχουμε ένα μεγαλύτερο ρυθμό, έχουμε ένα στόχο να πετύχουμε ένα καλύτερο στόχο μέχρι το 2020-2021. Και στο προσωπικό το 37% είναι γυναίκες ε, σε ό,τι αφορά τον κλάδο των μεταφορών. Και πάλι δεν έχουμε φτάσει στο 50% αλλά έχουμε στόχο να φτάσουμε εκεί. Και αν ε, μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι είμαι πολύ περήφανος ότι στην ε, μονάδα. Έχουμε ε, μία μονάδα στις υποδομές όπου η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είμαι πολύ περήφανος, πρόεδρος. Λοιπόν, ε, για να δούμε αν η επόμενη πρόεδρος της Παγκοσμίας Τράπεζας θα είναι γυναίκα για να έχουμε ίσες ευκαιρίες, αλλά να έχουμε ισότητα και στις αρμοδιότητες. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας, ευχαριστούμε κύριε Λιμπεράσκη για την εταιρική σχέση και ελπίζουμε να έχουμε την δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μου και θα έχουμε πάρα πολλά έργα που θα έρθουν, τη διασυνδεδεμένη κινητικότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα, όλες αυτές οι θεματικές. είναι μακροπρόθεσμες. Γιατί μπορώ να σας πω ότι μόνο με επενδύσει ε, στις υποδομές ε, αυτές ε, δεν αφορούν τα επόμενα 5-10 χρόνια, αλλά πρόκειται για ιδιαίτερα μακρόπνοα έργα. Και πρέπει να απαντήσουμε και στις παγκόσμιες προκλήσεις. Ευχαριστούμε πολύ του εκπροσώπου τη παγκόσμια Τράπεζας, μπορούμε να τους χειροκροτήσουμε. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Λιμπεράτσκι. Υπάρχει και ένα κοκτέιλ, αγαπητοί συνάδελφοι. Από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις 9, κάπω αργά. Αυτό θα γίνει στο σαλόνι ΑΣΠ, στο Ισόγειο. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Ξέρετε, όταν έχουμε ευθύνε, έχουμε και πολλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα και τα λέμε σε πολύ λίγο.